Συνάδελφοι, λέω να αρχίσουμε για να μην υπάρξει καθυστέρηση. Γιατί το απόγευμα είναι πολύ φορτωμένο. Πρώτα το σημείο 14 με βάση την έκθεση της Γιούτα Στάινμπροκ. έκθεση πρωτοβουλίας για αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασία ως στρατηγική βελτίωση των συνθηκών Εργασία στην Ευρώπη. Οι συντονιστές το είχαν προτείνει λόγω της σημασίας που παίρνει αυτό το θέμα σε ενωσιακό επίπεδο. Δεν είναι τίποτα καινούργιο, αλλά έχει προσλάβει νέες διαστάσεις και επικαιρότητα λόγω της μεγάλης αύξησης των διαμεθοριακών δοσοληψιών και την κατάσταση στις ηθικές εργασίας των λιγότερο προστατευμένων εργαζομένων. Είναι συζήτηση, είναι το θέμα αυτό σχετικό με την οδηγία για τις αποσπάσεις των εργαζομένων, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό. Έχει κάποια επικαιρότητα και λόγω του ότι οι επιθεωρήσεις εργασίας είναι αναποτελεσματικές λόγω των μέτρων λιτότητας και της μείωσης των δημοσίων δαπανών. Γι' αυτό λοιπόν οι συντονιστές δώσανε στη Γιούτα Στάινμπερκ την ευθύνη της ανάληψης αυτού, αυτής της έκθεσης. Και θα ακούσουμε τέσσερις εμπειρογνώμονες, μερικοί είναι ήδη γνωστοί στην Επιτροπή μας, γιατί τους έχουμε ξανακούσει. Ο Λούντο Μπέκ πρώτα, που είναι σύμβουλος στο Υπουργείο Εργασίας του Βελγίου, Φρανσουά Έγγελ σύμβουλος στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών του Λουξεμβούργου, Χάινς Φρίτς, που είναι υπεύθυνο για το τμήμα ασφαλείας στο Συνδικάτο Ίγκε Μετάλ της Γερμανίας και ο Κλόντε Μανουέλ Τριόμφ, που είναι από την επιθεώρηση εργασίας ο Ρόψος και που ονομάζεται Αστρέα. Σας ευχαριστώ και τους τέσσερις. Αλλά πριν σας δώσω το λόγο θα ζητήσω από την εισηγήτρια Γιούτα Στάινμπρουκ να μας παρουσιάσει το γενικότερο πηλέσιο της έκθεσής της και τα βασικά ερωτήματα που θα ήθελε να απαντήσετε. Ορίστε. Ε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το αναφέρατε ποια είναι οι λόγοι που η Επιτροπή μας ασχολείται με το θέμα αυτό των ελέγχων στην Ευρώπη. Ευχαριστώ τους εμπρογνώμονες που είναι σήμερα παρόντες, που ήρθαν εδώ για να μας δώσουν περισσότερες γνώσεις για το πώς έχει η κατάσταση, για το ποιες είναι οι προκλήσεις, πώς θα λειτουργήσει στο μέλλον όλο αυτό το σύστημα ελέγχων στην Ευρώπη εδώ στο Κοινοβούλιο ασχολούμαστε με το θέμα αυτό, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς και η Κομισιόν επίσης βρίσκεται σε μια φάση διαβούλευσης και ακριβώς με αυτό ασχολείται. Να υπάρξει δηλαδή μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα, η έλεγχη είναι ιδιαίτερως ε, σημαντική για, ε, για την απασχόληση για την ε, προστασία της, προ... της νόμιμης απασχόλησης, η οποία είναι πολύ σημαντική. Αυτές οι επιχειρήσεις θέλουν να κρατήσουν τους ε, εργαζόμενους τους, θέλουν να μπορούν να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό, όχι να πλήττονται από αυτό και γι' αυτό θα πρέπει να ε, μπορέσουμε να εμποδίσουμε την, τις παραβάσεις στο, των διαφόρων εργοδοτών. Επίσης η αδήλωτη εργασία είναι ένα σημαντικό θέμα. Φτάνει το 18,8% του ΑΕΠ. Και γι' αυτό υπάρχουν και χώρες που η ζημιά αυτή φτάνει και ακόμα το 30% του έπτους. Από τη μία λοιπόν έχουμε τελείως αδήλωτες δραστηριότητε, απ' την άλλη έχουμε και κάποιες εργασιακές σχέσεις όπου οι ε, εργοδότες ζητούν από τους εργαζόμενους να δουλέψουν κάποιες ώρες ή κάποιες μέρες τη βδομάδα και να δηλώσουν ότι δουλεύουν πλήρως. Ε, υπάρχουν επίσης, ε, υπάρχει κατάχρηση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στο χώρο εργασίας και πολλά ακόμη. Επίσης, υπάρχουν πολλές ε, συνέπειες, υπάρχει αντίκτυπο στους εργαζόμενους σε ό,τι αφορά την μετεκπαίδευσή τους, την κοινωνική τους ασφάλιση, τον, τον αποκλεισμό τους από την κοινωνία και από την άλλη μιλούμε και για την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και μιλούμε και για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Συνολικά, είπατε Πρόεδρε ότι αυτή η συζήτηση για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αποσπάσεις έδειξε ότι το, σημείο των, το θέμα των ελέγχων μάλλον είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, αρκετά αντικρουόμενο ζήτημα. Όλοι όμως συμφωνούμε ότι θέλουμε επι, ε, αποτελεσματικούς ελέγχους έτσι ώστε να, ε, να απαλείψουμε κάθε δυνατότητα ε, κατάχρησης, αλλά όλα τα κρατη λένε ότι θέλουν να εξοικονομήσουν ε, χρήματα και απ' την άλλη ξεχνούμε τις ε, τεράστια, τα τεράστια ποσά που χάνει το κάθε κράτο λόγω ακριβώ τη αδήλωτη εργασία. Σε πολλά κράτη-μέλη οι έλεγχοι, οι εργασιακοί πραγματικά ε, πάσχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό ακριβώ σε καιρό κρίση όπου οι δημόσιοι προπολογισμοί προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες ε, ε, ε, μειώσεις και περικοπές, τότε προκύπτουν περισσότερα προβλήματα. Υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες, αλλά αν δεν υπάρξει επιτόπου έλεγχος στα κράτη-μέλη, ό,τι και να λέει η οδηγία δεν ωφελεί. Και πέραν των, εργαζομένων και οι επιχειρήσεις πλήττονται και κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντιποκριθούν στον ανταγωνισμό. Μαύρη εργασία επίσης οδηγεί σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και πώς θα γίνει ε, όταν η Κομισιόν και ε, από τη μία δεν, από τη μία καταδικάζει την μαύρη εργασία αλλά δεν καταδικάζει το κοινωνικό ντάμπινγκ. Την επόμενη εβδομάδα θα υποβάλω εγώ την έκθεσή μου στην Επιτροπή μας. Δύο τμήματα θα έχει, καταρχάς το εθνικό επίπεδο και μετά την ευρωπαϊκή διάσταση. Εδώ μιλούμε για τις βασικές αρχές, ε, για εθνικούς αποτελεσματικούς ελέγχους. Πρέπει να δούμε ποιος ελέγχεται, πώς ελέγχουν οι αρχές, πώς θα πρέπει να είναι στελεχωμένες, ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές, θα υπάρξουν υποδείγματα σε ό,τι αφορά την συνεργασία μεταξύ αρχών. Και στο δεύτερο τμήμα θα μιλήσουμε με συστάσεις πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε ε, να υπάρξει καλύτερη ανταλλαγή διασυνοριακά των δεδομένων, ε, για ενίσχυση των ελέγχων διασυνοριακά, καθώς επίσης ε, και έλεγχο του κοινωνικού ντάμπινγκ στην Ευρώπη. Χαίρομαι που σήμερα είναι εδώ οι εμπειρογνώμονές μας, γιατί μπορούν να μας δώσουν πολύ καλές πληροφορίες, μπορούν να μας δώσουν την εμπειρία τους και χαίρομαι για τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και θα δώσω καταρχήν το λόγο στον κύριο Μπέκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Γενικά η αδήλωτη εργασία και η απάτη προσπασμένων εργαζομένων στην Ευρώπη παραμένει δύσκολο να μετρήθει. Αυτό θέτει δυσκολίε για όσου χαράζουν την πολιτική και ιδίω για τι επιθεωρήσει εργασία, καθώ προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο σε όλες τις πτυχέ του και να αναπτύξουν συγκεκριμένες πολιτικές και να βελτιώσουν τις επιθεωρήσεις τις πολιτικές ε, ή τουλάχιστον να παρακολουθούν ε, τέτοια φαινόμενα πάτης. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις στο να μειώσουν την αδήλωτη εργασία και να διασφαλίσουν ε, συνθήκες αξιοπρεπούς εργασίας για αυτούς τους εργαζομένους φαίνεται μέσα από την ανάγκη για κατευθυντηρίες γραμμές κοινή πολιτικής μεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Βέλγιο έχει θετική στάση απέναντι στις προτάσεις της Κομισιόν. Έχει, έχουν ανακοινωθεί οι προτάσεις αυτές εδώ και καιρό και υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες. Οι επιθεωρήσεις εργασίας αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες και προκλήσεις για να παρουσιάσουν αποτελέσματα στην καταπολέμηση της αδειλωτής εργασίας ε, και εργαζόμενοι και εργοδότες ε, συχνά δεν συνεργάζονται ε, γιατί οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους ή επειδή εργαζόμενοι στη μαύρη οικονομία δεν πληρώνουν φόρους ή για λόγους νόμου περιορισμού οι εργοδότες ε, θέλουν να μειώσουν το κόστος, ε, το λειτουργικό κόστος ε, και να αποφύγουν το όριο που επιβάλλεται από την νομοθεσία. Αυτό εξηγεί το πόσο σημαντική είναι η συνεργασία με τους παραδοσιακούς stakeholders όπως οι κοινωνικοί εταίροι, όπως και το ότι είναι σημαντικό να συνεργαστούμε με παρατηρητήρια, πανεπιστήμια, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα. Το Βέλγιο έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό συνεργασίας όπου συμμετέχουν και οι επιθεωρήσεις, ε, οι, κοινωνικοί, οι υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας ε, και οι 21 υπηρεσίες ε, συναντούνται μία φορά το μήνα υπό την Προεδρία του Δημόσιου Κατηγόρου η υπηρεσία οργανώνει δύο ημέρες πολυτομεακών επιθεωρήσεων από τις περιφερειακές ομάδες παρέμβασης ε, κάθε μήνα. Πρόσβαση στις πληροφορίες άλλων ιδρυμάτων βρίσκεται σε διάφορα στάδια ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμεση πρόσβαση, ηλεκτρονική ανταλλαγή μεταξύ των επιθεωρήσεων και άλλων σχετικών αρχών χρησιμοποιείται στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες για άντληση δεδομένων όμως εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα για άλλες χώρες κυρίως ό,τι αφορά τις φορολογικές αρχές. Το Βέλγιο έχει παράσχει μια καλή πρακτική, έχουμε ε, την ε, τράπεζα σταυροδρόμη για την κοινωνική ασφάλιση αποτελεί μια ομοσπονδιακή υπηρεσία με τριμερή διακυβέρνηση που δίνει πληροφορίε στι επιθεωρήσει για να σχεδιάσουν δράσει και να ερευνήσουν υποθέσει. Πάνω από 2.000 ιδρύματα και σε τοπικό επίπεδο ε, συνδέονται μεταξύ τους και πάνω από 722 εκατομμύρια μηνύματα ανταλλάχθηκαν το 2011 μέσω αυτής της πλατφόρμας. Κάθε ίδρυμα καταγράφει και επικαιροποιεί τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας. Τα προστατευμένα δεδομένα λόγω ιδιωτικότητας είναι προσβάσιμα μόνο για την κεντρική διαχειριστική αρχή. Οι ηλεκτρονικές αιτήσει είναι διαθέσιμες για τους εργοδότες, έροντας ε, το άχθος, το διοικητικό, όπως ε, το τιμόν άμεση δήλωση απασχόλησης για να εγγραφούν ε, νέοι απασχολούμενοι στο Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο Βέλγιο επιθεωρήσεις έχουν ε, μόνιμη πρόσβαση στον τιμώνα, δηλαδή σε αυτή την υπηρεσία δήλωσης ε, απασχόλησης στη Λιμόσα, βάση δεδομένων που αποτελεί ένα μέσο ελέγχου στην καταπολέμηση της απάτης και το θέμα του ανταγωνισμού δαπών εργαζομένων που δέχονται να εργαστούν με χαμηλότερους μισθούς ε, και δεν σέβονται τη βελγική νομοθεσία. Ένα άλλο σύστημα είναι το ΟΑΣΙΣ, Πρόκειται για μια υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης που έχει σχεδιαστεί για να καταπολεμήσει την απάτη στην κοινωνική ασφάλιση. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από το ΆΣΙΣ παρέχονται μέσω των ε, καναλιών ε, της ε, Τράπεζας Κοινωνικής Ασφάλισης που ανέφερα νωρίτερα. Η εφαρμογή αναλύει δείκτες απάτης όπως μη συνήθειά αύξηση ή μείωση του τζίρου και ξαφνική πρόσληψη απόλυση μεγάλου αριθμού εργαζομένων και ταξινομεί τη επιχειρήσεις σε επίπεδα κινδύνων. Ένα άλλο σύστημα είναι το Genesis, ε, το οποίο συλλέγει αποδείξεις από τις Εθνικές ε, Υπηρεσίες Επιθεώρησης αποτελεί ένα κοινό μητρό έρευνος με πρόσβαση στον Τιμόνα, στο Λιμόσα και σε άλλες βάσεις δεδομένου, και έτσι αποφεύγεται η επικάλυψη των επιθεωρήσεων από διάφορες αρχές. Το software επικαιροποιείται καθημερινά και συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για τις επιθεωρήσεις, τους λόγους για την επίσκεψη και τα αποτελέσματα. Ένα άλλο σύστημα είναι το DOLSIS, πρόκειται για μια νέα εφαρμογή, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2011 και επιτρέπει στους δημόσιους φορείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα κοινωνικής ασφάλισης. Η τράπεζα σταυρωτών των επιχειρήσεων, όπου εγγράφονται όλες οι επιχειρήσεις και οι οικονομικές μονάδες ε, με την ταυτοποίηση των ε, αρμοδίων. Επίσης, με αυτά τα μέσα έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις πληροφορίες επιπρόσθετα, μια συνεργασία. Μια συμφωνία συνεργασίας υπεγράφει μεταξύ των ε, εθνικών επιθεωρήσεων και των φορολογικών αρχών τον Ιανουάριο του 2010 για την ανταλλαγή πληροφοριών. Και αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση με τη Γαλλία για μια πιθανή άμεση πρόσβαση των αρχών και των δύο χωρών στα συστήματα πληροφοριών. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χρήση των κοινών πλατφόρμων, όπως είναι η KSS, Knowledge Sharing System, για την ασφάλεια και την υγεία, στο χώρο εργασίας δεν ε, ε, έχει αντιστοιχεί όταν μιλάμε για την αδήλωτη εργασία, κυρίως ε, επειδή των ορίων που τίθεται από την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ακόμη και αν ένα βήμα έχει γίνει ήδη με το σύστημα πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς για την μετάθεση των εργαζομένων, ε, μία δηλαδή εφαρμογή που επιτρέπει στις αρχές περιφερειακές και τοπικές αρχές να επικοινωνούν ε, μεταξύ τους ε, θέτοντας ερωτήσεις και απαντήσεις. Και αυτό λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2011. Στις 18 Φεβρουαρίου 2011 οι επεθεωρήσεις πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη χάρτα της Μπρίζ ε, προωθώντας την ε, προωθώντας ένα έγγραφο που κύρωνε την ανάγκη για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και της διασυνοριακής απάτης με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου υπάρχει μια πολλαπλή εντολή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, μάλλον, συγγνώμη, η επιθεώρηση αποτελεί με δημόσια λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργάζεται με τις φορολογικές αρχές ε, και με τις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλειας. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη να ε, προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ διάφορων φορέων όπως επιθεωρήσεις εργασίας και των φορολογικών αρχών προκειμένου να αποτραπούν τέτοιες απάτες. Το Βελγικό Υπουργείο Πασχόλησης δήλωσε την ικανοποίησή του που το project της οδηγίας επιβολής ενδυναμώνει τη δυνατότητα των κρατών μελών να διασφαλίσουν μια ορθή εφαρμογή της οδηγίας απόσπασης των εργαζομένων η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη καλύτερα αυτά τα μέσα έχει αυξηθεί προκειμένου να ενδυναμωθεί η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακόμη περισσότερο. Νομίζω ότι έχω υπερβεί και το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου. Για να ολοκληρώσω με ένα τελευταίο σχόλιο. Η πρόθεση ορισμένων κρατών μελών να παράσχουν ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στα κράτη-μέλη γενικά. Είναι επίσης ε, κάτι θετικό, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε για έναν ίσο μισθό για ταυτόσιμη εργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτά που είπατε, για την οδηγία για τις αποσπάσεις, η Επιτροπή μας έχει ψηφίσει με τρόπο σύμφωνο με αυτά που είπατε. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον επόμενο εμπειρογνώμονα τον Φρανσουά Ιγγέλ για τους βιοτέχνες του Λουξεμβούργου, θα ήθελα να καλωσορίσουμε εδώ μερικούς επισκέπτες από την εκλογική μου περιφέρεια υπό την ηγεσία του Δημάρχου Ίγκεμπουμ, ο Φραγκίσκος Έγγελς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πολύ που είμαι σε θέση εδώ να σας μιλήσω για τις επιθεωρήσεις εργασίας γιατί είναι ένα θέμα που με ενδιαφέρει πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Όταν εξετάζουμε τις επιθεωρήσεις εργασίας στις επιχειρήσεις διαπιστώνουμε ότι γίνονται με πολύ άσκημο τρόπο. Λόγω κυρίως του καταπιεστικού χαρακτήρα τους ενώ η νομοθεσία προβλέπει σε πολλές χώρες πολύ πιο ευρύ πεδίο εφαρμογής των ε, ελέγχων και προβλέπει οι επιθεωρήσεις της εργασίας να έχουν σαν στόχο τον έλεγχο και τις συμβουλές και ίσως και την τιμωρία των επιχειρήσεων. Αλλά αν δούμε με, ποιο, με ποια σειρά εφαρμόζονται οι δικαιοδοσίες αυτές, διαπιστώνουμε ότι καταρχήν γίνεται συμβουλή των επιχειρήσεων. Ενώ στην πράξη δεν ακολουθείται αυτή η λογική. Γιατί αυτό, γιατί. Θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω λιγάκι την άποψή μου για τις τρεις αυτές δικαιοδοσίες. Γιατί το Συμβούλιο δεν προώθησε περισσότερο τις επιθεωρήσεις εργασίας. Μάλλον γιατί στέλνουν ανίκανους ανθρώπους χωρίς προσόντα στις επιθεωρήσεις αυτές, ανθρώπους που δεν ξέρουν από δίκαιο, εργασιακό δίκαιο, για τα θέματα της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων δεν τους ενδιαφέρει έρχονται και λένε στις επιχειρήσεις δεν είναι καλά αυτά που κάνετε. Αν όμως η επιχείρηση ρωτήσει και τι μπορώ να κάνω, παντάνε «Α, αυτό δεν είναι δική μου δουλειά». Α, αυτο δεν ειναι δικη μου δουλεια α δεν τα κάνετε καλά. Πάντως σε πολλές επιθεωρήσεις, μερικές τουλάχιστον, έρχονται μηχανικοί που είναι πολύ, έχουν πολλά προσόντα και είναι γνώστες για τα θέματα της υγείας αλλά συνήθως είναι κλεισμένοι στο γραφείο τους και δεν πηγαίνουν επί τόπου ποτέ. Είπαμε ότι στόχος είναι να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την νομοθεσία που αφορά την, εργασία και ασφάλεια, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Τώρα για τους ίδιους τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις. Οι έλεγχοι λειτουργούν αρκετά καλά όταν είναι συγκεκριμένοι και ξαφνικοί δηλαδή για αεροδρόμια, για μεγάλες εγκαταστάσεις όπου η επιθεώρηση εργασία συνεργάζεται με την αστυνομία, το τελωνίο και κάνουν μια συγκεκριμένη επιχείρηση που τη βλέπουμε μετά και στις εφημερίδες. Αλλά αυτό που δεν λειτουργεί είναι ο έλεγχος των μικρών εγκαταστάσεων, η πρόσωψη του γείτονα το κτλ. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές και γι' αυτό δεν γίνονται και οι έλεγχοι, επιθεωρητές και επιθεωρήσεις. ούτε ελέγχουν για την παράνομη εργασία η οποία σημειώνεται συνήθως σε μικρές επιχειρήσεις. Τώρα για τις κυρώσεις που επιβάλλουν και τα πυρόστιμα. Είναι προφανές ότι οι κανόνες υπάρχουν για να εφαρμόζονται και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος δεν τους εφαρμόζει πρέπει να τύχει κύρωση, και μάλιστα υποδειγματική για να μην μπορέσει στο μέλλον να συνεχίσει να υποφελείται από την παρανομία. Δεν είμαι λοιπόν καθόλου κατά των κυρώσεων, αλλά πρέπει κατά πρώτο λόγο να πληροφορηθεί ο κόσμος, οι επιχειρήσεις, για να μπορέσουν να προσαρμοστούν και να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία. Και τώρα για να καταλήξω και να εξοικονομήσω χρόνο από το προηγούμενο. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχουν επιθεωρήσεις εργασίας που είναι, είναι, εταίροι των επιχειρήσεων και τους, τις συμβουλεύουν και ως προς το εργασιακό δίκαιο, ιδίως διαμεθοριακό, όσο και ως προς την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και πρέπει ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που εκπροσωπώ εδώ να έρχονται έμπειροι επιθεωρητές, να γνωρίζουν θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια και οι έλεγχοι χρειάζονται μεν αλλά πρέπει να αφορούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί εκεί γίνονται οι περισσότερες παραβιάσεις και παρανομίες και να υπάρχουν αποτελεσματικές κυρώσεις. Αν διαπιστωθεί ότι οι επιχειρήσεις, ή ορισμένοι εργαζόμενοι ή μερικοί δίθεν ανεξάρτητοι δεν σέβονται την νομοθεσία για την εργασία, την ασφάλεια και την υγεία, τότε πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις υποδειγματικές για να μην επαναλαμβάνεται η παρανομία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ο τρίτος εμπειρογνώμων είναι ο Χάιντς Φρίτς που είναι υπεύθυνο του Τμήματος Υγείας και Ασφαλείας στο Συνδικάτο Ίγκε Μετάλ της Γερμανίας. Ja, vielen Dank, Frau Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας προσκαλέσατε σε αυτή την ε, πολύ σημαντική ακρόαση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η ίδια εκπροσωπεί 2,3 εκατομμύρια ασφαλισμένους, εργαζόμενους. Έχει περίπου 300, οι οποίοι εργάζονται σε περίπου 300 ε, ξεχωριστές, ε, 300.000 ξεχωριστές επιχειρήσεις. Χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Υπάρχουν, ε, υπάρχει ένας πολύ μικρός αριθμός μεγάλων ε, επιχειρήσεων, μεγάλων εταιριών, με πολύ ψηλό με επίπεδο προστασίας που δεν θα χρειάζονταν οποιαδήποτε παρέμβαση, έχουν δική τους εμπειρογνωμοσύνη ε, και η εκπροσώπηση επίσης των εργαζομένων γίνεται στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Μετά, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός εταιριών οι οποίες έχουν ε, καλές προθέσεις, αλλά τους λείπει η εμπειρογνωμοσύνη. Όπου ο από την, ε, συνήθως ε, έχουν, υπάρχουν πολλές ε, γνώσεις από πλευράς μηχανικής κτλ. Αλλά σε ό,τι αφορά το διοικητικό άχθος, το, το, την καθημερινή εργασία των εργαζομένων δεν έχουν πολλές γνώσεις και εκεί παρεμβαίνει η γεμετάλ Και Επίσης αυτή που υπάρχει και ένας αριθμός ε, εταιριών που μας δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα, που ε, γνωρίζουν και ενσυνείδητα παραβιάζουν τη σχετική νομοθεσία. Το Οι έρευνες που κάναμε από το 2009 επιβεβαίωσαν αυτό που ούτως ή άλλως ξέραμε, ότι πολλοί χρησιμοποιούν ε, αυτή τη ε, δυνατότητα όταν ε, είναι νομικώς επιβεβλημένο. Σε άλλες χώρες βέβαια είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα, αλλά στη Γερμανία υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση από τους επιθεωρητές εργασίας. Πιο κάτω έχουμε λόγους όπως οι απαιτήσει των ε, πελατών κτλ. Η πίεση λοιπόν που κινεί τον, τον εργοδότη είναι μικρότερη για, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, αυτό συμβαίνει για διάφορους λόγους, αρκετά περίπλοκους. Η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ε, εφαρμόζεται στην ε, Γερμανία Βεβαίω ε, υπάρχουν πολλέ φορέ προβλήματα διότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία είναι αρκετά ασαφή πολλέ φορέ. Δηλαδή ακόμη και σε αυτού που έχουν τι καλέ προθέσει, μέχρι αυτού που ψάχνουν τα νομικά κενά, δημιουργούνται προβλήματα γιατί αυτός που έχει καλή πρόθεση δεν ξέρει τι ακριβώς να κάνει, επομένως έχει ελλείψεις, ξέρει την νομοθεσία αλλά δεν ξέρει ποιος μπορεί να τον βοηθήσει και ποια μέτρα πρέπει να πάρει και αυτός που έχει την πρόθεση να παραβιάσει τον νόμο ε, μπορεί να το κάνει. Γιατί υπάρχουν παράθυρα και πόρτες ανοιχτές. Μια που ακριβώς δεν είναι ε, συγκεκριμένη η νομοθεσία. Οι διατάξεις λοιπόν δεν είναι αρκετά ακριβείς έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε όλα αυτά τα παραθυράκια τα νομικά που υπάρχουν. Αυτό ισχύει για όλα τα είδη εργαζομένων. Βέβαια ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντα το σημείο αναφοράς ένας ε, κλάδος δεν μπορεί να, επειδή υπόκειται σε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, να μειώνει τα εργασιακά του πρότυπα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις. Όσο πιο συγκεκριμένες είναι οι διατάξεις, τόσο πιο εύκολο είναι να τις, να τις εφαρμόσουμε. Και τόσο πιο εύκολο είναι βεβαίω να δούμε και αν εφαρμόζονται και να ελέγξουμε αν εφαρμόζονται σωστά και να παρέμβουμε αν δεν εφαρμόζονται. Η ίδια είναι της άποψης ότι η νομοθεσία που υπάρχει έχει μεγάλες ελλείψεις σε ό,τι αφορά τις ε, ψυχικές ασθένειες. Ναι. Δεν αντικατοπτρίζεται αυτό πουθενά στην νομοθεσία. Και αυτό σημαίνει επιβάρυνση χωρίς όμως και η επιθεώρηση εργασίας ή ο εργοδότης να μπορεί να παρέμβει για να αλλάξει κάτι. Και τέλος, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, συνεκτικές οι διατάξεις που αφορούν τα εργασιακά θέματα. Υπάρχουν πάρα, πολλές, πάρα πολλοί ορισμοί οι οποίοι μπερδεύουν τόσο πολύ τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τηρήσουν την νομοθεσία. Mm και να εφαρμόσουν τις διατάξεις. Ε, και σαν να μην φτάνει αυτό, ένα από τα βασικά μας προβλήματα είναι ότι και στη Γερμανία το προσωπικό των, ε, ε, των επιθεωρήσεων εργασία είναι πάρα πολύ λίγο. Συνέκρινε εδώ τα δεδομένα από το 2002 στο 2011, 10 δηλαδή χρόνια αναφορών, και εδώ βλέπετε ότι το προσωπικό μειώθηκε σε όλα τα κρατήδια κατά 28%. Βεβαίω αυτό είναι το εργατικό δίκαιο, είναι θέμα κρατηδίου στην, στη Γερμανία, είναι ομοσπονδιακό κράτος η Γερμανία, αλλά κάθε κρατήδιο μείωσε το ε, προσωπικό του. Στην Βόρεια Ρινωνία Βεσφαλία ε, κράτησε 85 χρόνια μέχρι να φτάσει σε ένα σωστό επίπεδο η επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή μιλάμε για ανθρώπους ε, τρίτης γενιάς. Τώρα, η πίεση έχει να κάνει και με τις εταιρείε που επισκέπτονται οι επιθεωρητές. 120.000 ε, εταιρείε από 4 εκατομμύρια ελέγχθηκαν. Πολλές, αυτές, πολλές από αυτές επανειλημμένως. Βεβαίως υπάρχει μεγάλος, ε, είναι ε, εταιρείε υψηλού κινδύνου, αλλά αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να καλύψει η επιθεώρηση εργασίας όλες τις εταιρείες. μέσω ακριβώ ε, ε, των περικοπών στο, στις, ε, στους, ελεκτές, στους το πρόβλημα έχει οξυνθεί όπως λέει ένας από τους βασικούς μας εταίρους που μας έδωσε αυτά τα στοιχεία και δυστυχώς η δουλειά δεν, δεν μπορεί να γίνει, οι έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν αποτελεσματικά τότε που βεβαίω ε, δημοσιεύτηκε η έρευνα αυτή, τώρα ε, έτσι είχαν τα πράγματα. Βεβαίω ε, θα θέλαμε όλοι οι επιθεωρήσει εργασία να είναι περισσότερε, να, είναι, να δείτε περισσότερη προσοχή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρξουν σαφέστερες διατάξεις, να υπάρξουν σαφέστερες οδηγίες, τι είναι κυρώσιμο και κυρίως τι γίνεται και με το ψυχικό την ψυχική πίεση που υπάρχει. Αυτά από μένα ευχαριστώ. Merci. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής είναι ο κύριος Κλόντε Μανουέλ Τριόμφ, ο οποίος είναι διευθυντής της Ένωσης Τραβαγιαν Employee Ρουψοσιετέ και υπενθυμίζω ότι είχαμε ξανασυζητήσει μαζί του όταν ε, εξετάσαμε την έκθεση ΣΕΡΚΑΣ ε, για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές. Ε, όχι απλώς είμαι διευθυντής αυτής της Ένωσης στη Γαλλία αλλά μεταξύ των τεσσάρων ομιλητών είμαι ο μόνος επιθεωρητής γιατί στο πρώτο στάδιο, στο πρώτο τμήμα της επαγγελματική μου σταδιοδρομίας ασχολούμαι με το θέμα αυτό, αλλά ήμουν και πρόεδρος της Γαλλικής Ένωσης Επιθεωρητών Εργασίας και τα τελευταία έτη έχω ασχοληθεί με project είτε από το όνομα του ε, Εθνικού Γραφείου και στις τρεις βαλτικές χώρες αλλά έχω ασχοληθεί και με project που έχουν να κάνουν με την απόσπαση των εργαζομένων και με τη συνεργασία μεταξύ των δημοσίων αρχών και των επιθεωρήσεων εργασία. Δεν θα σας μιλήσω λοιπόν για το γαλλικό σύστημα επιθεώρησης εργασίας αλλά θα σας μιλήσω για ένα κίνδυνο που κατά την άποψή μου είναι σημαντικό σε ό,τι αφορά το σύστημα σύνολο των συστημάτων επιθεώρησης εργασίας στην Ευρώπη. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να υπενθυμίσουμε είναι ότι πως όταν μιλάμε για επιθεώρηση εργασίας, καταρχήν ε, οι όροι αναφοράς μας δίνονται από το Γραφείο Επιθεώρησης Εργασίας και από τη Σύμβαση 81 που έχει κυρωθεί από τα 28 κράτη-μέλη της Ένωσης. Επομένως, οι όροι αναφοράς ε, προέρχονται από μια παγκόσμια οργάνωση. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ευρωπαϊκοί τέτοιοι όροι ε, τέτοια συγγραφή υποχρεώσεων, τέτοια συγγραφή υποχρεώσεων, όμως ε, να σας πω ότι πίσω από αυτό το ίδιο όνομα υπάρχουν πολλές διαφορετικές πραγματικότητες. Υπάρχουν ε, πολλές αποχρώσεις στην εικόνα, αλλά έχουμε γενικά δύο μεγάλες κατηγορίες συστημάτων στην Ευρώπη, μαζί και με κάποια ενδιάμεσα βεβαίω συστήματα. Θα έλεγα ότι αυτά τα δύο συστήματα, γκροσομόντο, αφορούν ε, περίπου το 50% των ευρωπαϊκών κρατών. Ε, δηλαδή, το ένα σύστημα εφαρμόζεται στο νότο και ανατολικά, νότια του Βελγίου, ενώ το άλλο σύστημα εφαρμόζεται στις βόρειες και στις βορειοανατολικές χώρες της Ευρώπης. Τώρα, το πρώτο σύστημα που αποκαλείται επιθεώρηση εργασίας ή των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ένα γενικό σύστημα, δηλαδή ασχολείται με μια σειρά σχέσεων εργασίας, φυσικά με το θέμα της ε, υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, αλλά και με τους μισθούς, με την ε, παράνομη εργασία κτλ. Έτσι, λοιπόν, ε, το σύστημα αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα σύστημα γενικό, να το χαρακτηρίσουμε σε ένα γενικό σύστημα. Οι επαγγελματίες ε, προέρχονται συνήθως από διάφορους ε, κλάδους, έχουμε πολλούς νομικούς, οικονομολόγους, ανθρώπους που έχουν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Τώρα το δεύτερο σύστημα ασχολείται όχι αποκλειστικά αλλά ουσιαστικά ασχολείται με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και σπανίως ονομάζεται επιθεώρηση εργασίας στην Ευρώπη. Μιλάμε για αρχή υγείας και ασφάλειας ε, στο χώρο εργασίας. Ε, δεν πρόκειται για το ίδιο και υπάρχουν κάποιες σημασιολογικές διαφορές που είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί καθορίζουν και τις αρμοδιότητες ε, των ανθρώπων. Και σε αυτό το δεύτερο σύστημα έχουμε κυρίως εμπειρογνώμονες στο θέμα της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Τώρα, κάτι άλλο που πρέπει να δούμε όταν μιλάμε για το θέμα αυτό στην Ευρώπη ε, για την επιθεώρηση πρόκειται για ένα σύστημα που δεν καλύπτει παρά τον ιδιωτικό τομέα, ενώ άλλο σύστημα καλύπτει και το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και ουσιαστικά έχουμε σύστημα διοικητικών κυρώσεων, ε, τα περισσότερα όμως είναι υπό την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, με εξαίρεση στην Πολωνία, όπου εκεί την αρμοδιότητα την έχει απευθεία στο Κοινοβούλιο. Επίσης έχουμε πολλά συστήματα αρχικής κατάρτισης και θα αναφερθώ στο γεγονός ότι ο τίτλος της ακρόασής σας λέει συνθήκες εργασίας και αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας. Όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν βρισκόμαστε εδώ στο θέμα των εργασιακών συνθήκων ε, της Ευρώπης Working Condition. Μιλάμε για Occupational Health and Safety, επαγγελματική υγεία και ασφάλεια. Και αν δείτε πώς η Eurofound ορίζει τις Working Conditions, τις συνθήκες εργασίας, έχουμε ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Όμω, ο τομέα των κοινών ορμοδιοτήτων, των επιθεωρήσεων εργασία δεν είναι οι συνθήκε εργασία, αλλά επαγγελματική υγεία και ασφάλεια και εγώ νομίζω ότι αυτό έχει πολλέ συνέπειε για το πώ συνεργαζόμαστε και λειτουργούμε από κοινού. Και ήθελα τώρα να θέσω μια ερώτηση. Σήμερα υπάρχει ένα είδος ολοκληρωμένου συστήματος στην Ευρώπη. Να έχουμε κάτι που το λέμε SLEEK, Senior Labor Inspectors Committee, που αποτελεί μια δομή αρκετά soft θα έλεγα και ουσιαστικά ασχολείται με την ανταλλαγή μεταξύ υπεύθυνων επιθεωρητών εργασίας οι οποίοι προσπαθούν να, να υλοποιήσουν κοινέ εκστρατείε για το θέμα της επαγγελματική υγείας και ασφάλειας και λίγο έχουν εργαστεί για τα μεθοδολογικά ζητήματα. Αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό στην Ευρώπη. Υπογραμμίζω ότι υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που συνεργάζονται τα συστήματα. Έχω κατά νου αυτά τα ευρωπαϊκά project για το θέμα τη απόσπαση των εργαζομένων και πολλέ διασυνοριακέ πρωτοβουλίε όπου οι χώρες από τις δύο πλευρές των συνόρων ε, ανταλλάσσουν πληροφορίες και κατόπιν υπάρχει και ένα δίκτυο των σχολών κατάρτισης ε, των επιθεωρητών. Αυτό είναι σημαντικό γιατί αυτό το σύστημα δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες, αυτό το σύστημα των σχολών. Θα ήθελα τώρα να προσεγγίσω τις κυρίες προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουν τα συστήματα επιθεώρησης εργασίας στην Ευρώπη. Καταρχήν, Πρόεδρε, είναι η μεταμόρφωση των επιχειρήσεων. Σήμερα ζούμε σε ένα πολύ παγκοσμιοποιημένο κόσμο με μια πολύ μεγάλη επιρροή των ε, δικτύων επιχειρήσεων και των ομίλων. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο όπου η υπεργολαβία, η συνεργολαβία και η εξωτερική ανάθεση έχουν ε, πολύ μεγάλο ρόλο. Δεύτερον, έχουμε διεθνοποίηση των αγορών εργασίας, αρκετά μεγάλη και μεγάλη ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόβλημα είναι πώς τα συστήματα αυτά λαμβάνουν υπόψη αυτή την ε, μεταμόρφωση και τελικά τι γίνεται στην πραγματικότητα. Και θα έλεγα ότι ένα από τα προβλήματα, και το υπογράμμισαν και άλλοι συνάδελφοι, πιστεύω ότι αφενό ο πληθυσμό των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αφήνεται κατά μέρο για μια σειρά λόγων που θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στη συζήτηση, αλλά επίση και το θέμα τη επιρροή των πολυεθνικών. Δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η τροποποίηση των κανόνων ε, του ε, της εργατικής νομοθεσίας. Μιλήσαμε πολύ για την ε, τροποποίηση των συμβάσεων για την εμφάνιση ελεύθερων επαγγελματιών, για την παράνομη εργασία, αλλά υπάρχουν λένε και περισσότερο ιδιωτικά πρότυπα, πρότυπα τα οποία ε, μπορεί να δημιουργούνται από τους κοινωνικούς εταίρους ε, στον τομέα της δραστηριότητας των στην επιθεωρήση αλλά δεν έχει αρμοδιότητα και επιθεωρήση εργασία, επειδή δεν επίπτουν αυτά στο νομικό σύστημα. Η ερώτηση είναι λοιπόν, ποια είναι αυτά τα νέα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιθεωρήσεις εργασία για να δράσουν και τι είδου κυρώσει μπορούν στο μέλλον να επιβάλλουν και ποια είναι η συμπληρωματικότητα μεταξύ των φορέων. Και θα ήθελα να κλείσω με κάποια σχόλια σε σχέση με, το, ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα. Καταρχήν, ναι, Υπάρχει αντικειμενικό ενδιαφέρον να έχουμε ένα τέτοιο πιο ολοκληρωμένο σύστημα. Έχουμε την κινητικότητα των εργαζομένων, έχουμε όλο ένα και περισσότερα είδη συμβάσεων, έχουμε το ρόλο κλειδί των πολυεθνικών και των ομοιόμορφων προτύπων μεταξύ των διαφόρων χωρών και κάποιες κοινωνικονομικές αλλαγές. Όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη. Όμως απέναντι σε όλα αυτά τα συστήματα επιθεώρησης εργασίας είναι εντελώς κατακαιρματισμένα στην Ευρώπη. Παραμένουν επικεντρωμένα σε εθνικές προσεγγίσεις ε, και στο περιθώριο των εξελίξεων. Παραδείγματο χάρη, ο Γερμανός συνάδελφος αναφέρθηκε στο θέμα των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Τα συστήματα επιθεώρηση εργασία, σίγουρα θα έλθουν να διαδραματίσουν ρόλο πολύ αργότερα από τους ε, υπόλοιπου φορεί. Και θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι ναι, σήμερα χρειαζόμαστε μια διασταυρούμενη δράση, αλλά χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από το σλικ, χρειαζόμαστε βάσεις δεδομένων και πραγματικά μοντέλα κατάρτισης. Υπάρχουν ήδη κάποιες πλατφόρμες ανταλλαγής πληροφοριών που πρέπει να αναπτυχθούν πολύ περισσότερο, γιατί σήμερα είναι αρκετά γραφειοκρατικές. Και ας μην μείνουμε στο θέμα των με μεταθέσεων των εργαζομένων, αλλά ας δούμε και άλλα ζητήματα, να δούμε και συστήματα μεθοδολογίας και συστήματα επιβολής κυρώσεων. Καθώς τα περισσότερα συστήματα επιθεωρήσης εργασίας ε, Παραδείγματο χάρη, στα περισσότερα συστήματα, όπως στη Γαλλία, το 1% είναι οι κυρώσει. Και αν ε, οι κυρώσει σήμερα δεν είναι αποτελεσματικέ και έχω κατά νου τις μεγάλες επιχειρήσεις και τα πολύπλοκα κέντρα λήψη αποφάσεων, ε, αν θέλετε, δεν κάνουμε τίποτα. Είμαστε μια σταγόνα στον ωκεανό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μάλιστα καταφέρατε να περάσετε και το χρόνο αγόρευσης χωρίς να σας διακόψω. Μπράβο σας. Και είπατε, παίρνοντα χάρη, ότι οι επιθεωρητέ εργασία οι τελευταίοι είδαν τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα και μπορώ να σα πω ότι εκεί και αξιολόγηση ήταν οι τελευταίοι που είδαν την υποβάθμιση ε, των δανείων για υποθήκες. Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο καταρχήν στην κυρία Λάμπερτς. Παρακαλώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Όλοι μας θεωρώ ότι, είναι, ότι πιστεύουμε πολύ, ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Όντως υπάρχει έλλειψη στον αριθμό επιθεωρητών εργασίας. Βέβαια αυτό δεν μας εκπλήσει γιατί όταν ε, πηγαίνουμε σε διάφορα επισκε... Ε, ταξίδια για να επισκεφτούμε διάφορες χώρες, ε, πάντα μας λένε ότι είναι πολύ, μικρο, πολύ μικρός ο αριθμός, πάντα ρωτούμε τι είδους σύστημα έχουν για τις επιθεωρήσεις εργασίας και πάντα μας λένε πολύ μικρά νούμερα. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και επίσης πρέπει να δούμε το, τους στόχους που θέτουμε, να συνεργαστούμε με τομείς που ίσως είναι πιο πολύ σε κίνδυνο, είτε είναι στην γεωργία, στην κατασκευή. Θα ήθελα τα σχόλιά σας για το αν πιστεύουμε ότι αυτό θα ήταν ένας αποτελεσματικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις, αυτούς τους λίγους πόρους που έχουμε. Ε, μπορώ να μαντέψω την απάντηση, αλλά αν μπορείτε απαντήστε μου. Σε ό,τι αφορά την ε, συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που μας ε, λένε συχνά όταν προσπαθούμε αυτό να το περάσουμε στην νομοθεσία, είναι ότι είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και δεν μπορεί να γίνει, όλα είναι διαφορετικά. Και αυτό ακούγεται σαν δικαιολογία, όχι σαν λόγος για να μην γίνει. Οπότε τι είδους στήριξη θα μπορούσε να δοθεί. Ε, το θέμα είναι ο χώρος για να υπάρξει, να οργανωθούν οι ε, πόροι. Τι ακριβώς φταίει και δεν μπορεί να υπάρξει συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Jsem rád, že se o problému inspekcí konečně začalo mluvit. Ale připrav που ξεκινήσαμε επιτέλους να μιλούμε για τις επιθεωρήσεις εργασίας. Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όταν ξεκινούμε να πάρουμε οποιαδήποτε μέτρα που θα μας οδηγήσουν σε ενοποιημένη εργασιακή νομοθεσία, όλα τα κρατημέλη αρχίζουν και μιλούν για τις παραδόσεις τους, για την ε, επικουρικότητα. Εγώ έχω εργαστεί ως ε, επιθεωρητής εργασίας. Όντως είναι πολύ ανασφαλής ε, η εργασία πια, η αγορά εργασίας γίνεται όλο και πιο ευέλικτη σε εισαγωγικά και όλα αυτά προφανώς είναι πολύ αντιπαραγωγικά σε σχέση με τα όσα αναφέρατε εσείς κύριοι. Η λύση είναι απλή, όπως είπε και η κυρία Λάμπερτς. Πόσους ε, επιθεωρητές εργασίας έχουμε, πόσοι υπάρχουν στα διάφορα κράτη-μέλη. Φανταστείτε πόσοι εργάζονται παράνομα στις διάφορες κατασκευαστικές, ε, σε διάφορα κατασκευαστικά ε, σημεία στις, ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Συνήθως ο μηχανικός είναι ο επιθετικός, αλλά πολλές φορές και οι εργαζόμενοι εκεί είναι πολύ επιθετικοί. Ελπίζω βέβαια τα πράγματα να μην καταλήξουν όπως καταλήγουν πάντα. Και κλείνοντας, να πω κάτι. Πρέπει να κάνουμε... Θέλουμε να κάνουμε πάντα το καλύτερο, αλλά συνήθως το αποτέλεσμα είναι κακό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με το επεξηγηματικό σημείωμα που έχουμε στην ε, έκθεση. Εκεί λέμε ότι αυτές, αυτές οι επιθεωρήσεις εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μαύρη εργασία. Οι ε, επιθεωρητές εργασίας πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν το θέμα της μαύρης εργασίας. Μιλήσατε πολύ για την προστασία των εργαζομένων κτλ. Όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη μαύρη εργασία. Γιατί εκεί πραγματικά υπάρχουν τεράστια ε, συμφέροντα. Ε, επίσης, Ε, το θέμα δεν είναι να είναι μόνο το γραφείο στη σωστό ύψος του εργαζόμενου κτλ. Το θέμα είναι να μπούμε στον πυρήνα του προβλήματος, να δούμε τι γίνεται και με την ηχορύπανση κτλ. Ε, τώρα, για τον κύριο Τριών. Μιλήσατε για το θέμα της προστασίας εργασίας και των επιθεωρήσεων εργασίας. Πολύ σημαντικό που το είπατε και που το διαχωρίζετε, αλλά νομίζω ότι ε, ο δεύτερος ομιλητής, ο κύριος Έγγελς, μίλησε κυρίως για τα καθήκοντα και των ε, επιθεωρητών αλλά και των μηχανικών κτλ. Νομίζω ότι εδώ βρισκόμαστε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι, ποια είναι αυτά τα βασικά καθήκοντα. Θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την, μαύρη εργασία, θέλουμε να απλώς να ε, διασφαλίσουμε την ε, νόμιμη εργασία, τι θέλουμε να κάνουμε το μας Φιλμπενιό και δυστυχώς ο κύριος Μπουλάν που είναι σκιώδης ε, του ΕΛΚ Δεν ξέρω, θέλετε να σας βάλω στον κατάλογο, γιατί διαφορετικά θα έχουμε κάποιον από το ΕΛ και το μας Χάντελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τέσσερις παρατηρήσει έχω που θέλω να καταθέσω. Ερώτημα προς τον κύριο Έγγελς, καταρχάς ε, όντως οι κανόνες ε, και η συζήτηση είναι πολύ σημαντική. Η συζήτηση πήγε κυρίως γύρω από, την, ε, ε, από τις Μιλούμε για κανόνες οι οποίοι τελικά δεν μας βοηθούν σε τίποτα, μένουν στο χαρτί, γιατί δεν υπάρχουν έλεγχοι που να γίνονται από τα κράτη-μέλη. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Το θέμα δεν είναι να μιλούμε για την προστασία της εργασίας, για την διασφάλιση της ε, ασφάλειας στην εργασία. Το θέμα είναι να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές που ακολουθούνται. Εγώ είμαι της άποψης ότι τα περασμένα χρόνια υπήρξε πολύ μεγάλη αύξηση ε, ψυχικού βάρους, ε, ψυχικής πίεσης όσο διαφορά τον, τους ελεγκτές και το τι πρέπει να ελέγξουν. Όπως ε, ε, συνέβαινε και με τους επιθεωρητές το 1830 στη Βρετανία. Κάτι άλλο που επίσης ήθελα να πω. Νομίζω ότι εδώ σε αυτή την δήλωση της Επιτροπής μας θα πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα της ευθύνης των επιχειρήσεων, των εταιριών. Πολλές φορές είναι συστηματική η παραβίαση των ε, δικαιωμάτων ε, των εργαζομένων. Ε, συνήθως παραβλέπουν οι εργαδότες όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, κάνουν πολύ επισφαλείς συμφωνίες. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει ένας, ε, ένας τρόπος να ελέγξουμε αυτή την κατάσταση. Επίσης, αν δεν υπάρξει νέα οργάνωση, τι θα γίνει. Στη Βαβαρία, και νομίζω ότι δεν είναι μόνο στη Βαβαρία, αλλά και αλλού, υπάρχουν ε, και κάποιες, ε, ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι επιθεωρητές εργασίας. Εγώ κάποια στιγμή πήγα incognito σε μια τέτοια επιθεώρηση και είδα ότι ο ε, ελεγκτής ε, είπε έτσι πολύ ντροπαλά ότι θα πρέπει να ελέγξει, ο επιθεωρητής είπε πολύ ντροπαλά ότι θα πρέπει να ελέγξει κάτι παραπάνω. Θα πρέπει λοιπόν κάπως να αλλάξουν τα πράγματα. Και τελευταία παρατήρηση σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Έγγελς για, τους, ε, για τις επιθεωρήσεις ελέγχων ε, και για τα tips, τις συμβουλές που πρέπει να δίνονται στις επιχειρήσεις για το πώς ε, λειτουργούν τα πράγματα αλλού. Ίσως εγώ να κατάλαβα λάθος. Αλλά αν εγώ πάω με το αυτοκίνητό μου στην εταιρεία για, ε, για έλεγχο και υπάρξει πρόβλημα με το αυτοκίνητό μου, το θέμα μου είναι αν θα μπορέσω να το διορθώσω. Όχι, ότι όχι να μου διαπιστώσει ο ότι έχω πρόβλημα, προφανώς. Οι συμβουλέ λοιπόν που δίνονται και οι κατευθυντέρε γραμμές θα πρέπει να βελτιώνουν την κατάσταση. Αν τώρα χρειάζονται οι εταιρείε συμβουλές για την αντιμετώπιση των ε, ατυχημάτων κτλ. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά Ινστιτούτα, αρκετά, ε, αρκετές σχολές που μπορούν να, να παράσχουν τέτοια πληροφόρηση. Ευχαριστώ κύριος ε, Μπενιόν και να ξαναδώσουμε το λόγο στην συγγετρία κύριος Μπενιόν. Ευχαριστώ να κάνω κάποια σχόλια. Σίγουρα δεν έχω κάποια ισχυρή άποψη σε σχέση με το ολοκληρωμένο σύστημα. Λειτουργεί καλύτερα από ένα σύστημα ειδικών, όμως τα συστήματα ειδικών ε, δεν ασχολούνται μόνο με την ασφάλεια και την υγεία. Και αυτό μου το δήλωσε τόσο επικοινωνία για την αδειλία του εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, έχουμε ένα σύστημα ε, όπου και η φορολογική υπηρεσία και η τελειωνική υπηρεσία έχουν αρμοδιότητες για την καταπολέμηση της αδειλωτής εργασίας, ε, γιατί φυσικά αν μιλάμε για αδειλωτή εργασία δεν καταβάλλονται και φόροι. Επίσης έχουμε και μία σειρά άλλων λειτουργιών, όμως ένα τμήμα της επιθεώρησης εργασίας ε, περνάει από το HMRC Έχουμε βέβαια και την, περιβαλλοντική, την υπηρεσία περιβαλλοντικής υγείας που διερευνά οποιαδήποτε περιστατικά σε εργοστάσια που μπορεί να έχουν αντίκτυπο στο περιβάλλον. Και ξέρετε για την υπηρεσία επαγγελματική υγείας και ασφάλειας. Επομένως, το θέμα είναι ότι οποιοδήποτε σύστημα κι αν έχει κανείς, είτε έχει ολοκληρωμένο σύστημα, είτε διάφορους οργανισμούς που στελεχώνονται από εμπειρογνώμονες, ακόμη και σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, θα χρειαστεί στους εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς. Νομίζω ότι και τα δύο συστήματα αυτή τη στιγμή υποφέρουν από έλλειψη σε προσωπικό και σίγουρα ε, υπάρχει δυσκολία να καταπολεμηθεί η αδηλωτή εργασία και η φοροδιαφυγή. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει τώρα να συζητήσουμε ιδιαίτερα το αν είναι ολοκληρωμένα τα συστήματα ή όχι και ε, αν καλύπτουν τις ανάγκες νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε είτε το ένα είτε το άλλο σύστημα αλλά πολλές φορές το πρόβλημα αφορά τους πόρους. Euh, Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας θέλω να ευχαριστήσω τους τέσσερις εμπειρογνώμονες. Στην Επιτροπή μας συζητούμε το θέμα αυτό από πολύ καιρό, από τότε που εγκρίναμε την έκθεση πρωτοβουλίας για την ανανέωση της στρατηγικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Όχι ότι θέλαμε να παρέμβουμε στη δουλειά των επιθεωρητών, αλλά να καθορίσουμε υψηλά πρότυπα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα λαμβάνοντας υπόψη τις ψυχοσωματικές ασθένειες, το άγχος κλπ. Θα ήθελα να ξαναρωτήσω όμως τους εμπειρογνώμονες κάτι για τις μεγάλες επιχειρήσεις εταιρείες είπατε ότι το καινούργιο και πιο δύσκολο καθήκον των επιθεωρητών είναι να πηγαίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλπ. Αλλά εγώ με την εισηγήτρια αρχίσαμε να σκεφτόμαστε ότι τα σκεφτήκαμε όλα αυτά για πρώτη φορά όταν επισκεφθήκαμε μια μεγάλη εταιρεία όπου η επιθεώρηση της εργασίας ήταν πιο δύσκολη λόγω των πολλαπλών αποσπάσεων των εργαζομένων. Γιατί επιθεωρεί κανείς τις συνθήκες εργασίας τοπικά, την υγεία, την υγιεινή, τη... λοιπά Αλλά μπορεί να υπάρχουν και θέματα πληρωμής ή των εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση και έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος το κατά πόσον πληρώνεται η εισφορά είναι και αυτό ένα θέμα. Και γι' αυτό η εντύπωση που αποκομίσαμε από την επίσκεψη εκείνη ήταν ότι πέρα από το Senior Inspection Labor Committee θα επανέλθω στην τελευταία φράση των διαφανειών του κυρίου Τριόμφ μπορεί ένα θέμα να είναι και η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Σώματος Επιθεωρητών, ίσως όχι αύριο, αλλά να. Δεν λέω να εξευρωπαϊστούν τα πάντα. Κάθε επιθεώρηση εθνική θα έχει τις ευθύνες της, αλλά αν υπάρχουν διαμεθοριακές διαφορές και ε, είναι αρμόδιες πολλαπλές ε, επιθεωρήσεις τότε ίσως να χρειάζεται κάποιος κοινό παρονομαστής όπως υπάρχουν φορολογικές δημιουργίες να υπάρξει και μια τέτοια δημιουργία ελίτ που να παρεμβαίνει όταν γίνονται τέτοιες παραβιάσεις που αφορούν πολλά εθνικά συστήματα δικαίου, πολλαπλά. Κάτι ανάλογο συζητήσαμε και για τη φοροδιαφυγή και για την καταπολέμηση των, της μόλυνσης στις ακτές. Είναι εδώ ολόκληρο κίνημα, τάση που νομίζω ότι μπορεί να ληφθεί υπόψη και στην επιθεώρηση εργασίας. Και τώρα δίνω το λόγο στην εισηγήτρια Ούτα Στάινμποκ. Ja, vielen Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω κάποια ερωτήματα κι εγώ για τους εμπειρογνώμονες, για τον κύριο Μπέκ. Αν έχω σωστή πληροφόρηση, το δικαστήριο ήταν, ε, έβγαλε απόφαση αντίθετη με το σύστημα λιμόζα, καταδίκασε το σύστημα λιμόζα. Ε, εμείς έχουμε συζητήσει και το ακούσαμε σήμερα και από τους εμπειρογνώμονες. Εσείς πώς το, πώς το αξιολογείτε αυτό. Υπάρχουν δυνατότητες ε, παρέμβασης και η, ε, ο αντίκτυπος ποιος είναι για το Βέλγιο. Η διασυνοριακή τώρα ανταλλαγή δεδομένων. Το άκουσα από πολλές πλευρές να λέγεται, η οποία είναι πάρα πολύ ελλειπής ε, και εντός της ε, Ευρώπης ε, τα κράτη-μέλη τελειώνουν τους ελέγχους μέχρι εκεί που φτάνουν τα σύνορά τους. Από εκεί και πέρα είναι απελπιστική η κατάσταση. Δεν δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες στα υπόλοιπα κράτη-μέλη, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει αυτή η χάρτα, είπατε, που ε, οι επιθεωρητές εργασίας από 11 χώρες υπέγραψαν. Αυτή η χάρτα έχει οδηγήσει σε κάτι συγκεκριμένο, έχει οδηγήσει σε κάτι θετικό, σε κάποια θετική αλλαγή, είχε κάποιες συνέπειες. Κύριε Έγγελς, είπατε ότι λείπει εκπαίδευση και αρμοδιότητες. Συνήθως ε, μιλούμε ε, για το βάρος που έχουν οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως όταν μιλούμε για προστασία στην εργασία. Αλλά κατά την άποψή σας είναι απαραίτητο να υπάρξουν ευρωπαϊκές διατάξεις ως προς αυτό για, ε, για να υπάρξει περαιτέρω εκπαίδευση των επιθεωρητών ή για το ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων. Πρέπει αυτό να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επίσης, μιλήσατε για το θέμα των επιθεωρήσεων σε μικρά ε, εταιρείε για, κατασκευαστικές, για κατασκευές. Κατά την άποψή σας αυτό πώς θα γίνει. γιατί και εκεί μπορεί να υπάρξει αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας, πώς μπορούμε να κάνουμε και ελέγχους επιθεωρής εργασίας και να, προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Νομίζω ότι και τα δύο σημεία είναι πολύ σημαντικά. Μετά, ένα ερώτημα για τον κύριο Φρίτς. Μιλήσατε για την προστασία της υγείας η οποία πρέπει να ασχοληθεί κυρίως με την ε, ψυχική επιβάρυνση. Έχετε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ή έχετε μια εικόνα για το πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η δική μας η ε, υπηρεσία στον Μπιλμπάο ασχολείται πολύ με το θέμα της πρόληψης. Πώς μπορούμε να το δούμε αυτό από την πλευρά της ε, επιθεώρησης εργασίας πάντα. Και για τον κύριο Τριόμφ, καταλαβαίνω αυτό που λέτε, Συμφωνείτε μαζί μου, έχω μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκές επιθεωρήσεις με την υποχρέωση ε, αυτό να είναι ένα ε, ευρωπαϊκό σύστημα. Ε, κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Μάλιστα δεν ε, θα έχετε μισή ώρα στη διάθεσή σας για να απαντήσετε ακόμη και αν δεν χρειάζεται. Θα έχετε πέντε λεπτά. Ο κύριο Λουδομπέκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να απαντήσω στι ερωτήσεις, να πω καταρχήν ότι πράγματι είχαμε μία απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για ένα τμήμα του συστήματος Λιμόσα. Ζητήσαμε κάποιους ορισμούς ε, σε σχέση με το να μπορούν να έρθουν ανεξάρτητοι εργαζόμενοι στο Βέλγιο και η απόφαση ήταν ότι ζητήσαμε πάρα πολλά και ότι ήδη είχαμε προσαρμόσει τη βελγική νομοθεσία και για τους ε, ανθρώπους ε, που είχαν αποσπαστεί στο Βέλγιο ήταν σχετική αυτή η απόφαση. Για μας ως επιθεωρήση εργασίας είναι σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή τη δήλωση, να έχουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουμε την απάτη στον τομέα αυτό και κυρίως την απάτη σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίε. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. είχε να κάνει με το ότι οι επιθεωρήσεις ε, σταματούν, περιορίζουν μάλλον ε, τη δράση τους ε, στα περιφερειακά σύνορα. Γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε πολλές καλές πληροφορίες και συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και μέσω διμερών συμφωνιών. Ακόμη και μέσω τέτοιων συμφωνιών προσπαθούμε να προβούμε σε ανταλλαγή πληροφοριών και γι' αυτό σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα ανταλλαγή πληροφοριών από το οποίο να υποφελούνται όλες οι χώρες. Εγώ δεν πιστεύω σε ένα γενικευμένο σύστημα, αλλά πιστεύω σε μία επιθεώρηση με εξειδικευμένες μονάδες που όμως θα επικοινωνούν καλά μεταξύ τους οι μονάδες αυτές και θα βάζουν και στο ίντερνετ όλες τις πληροφορίες. Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με ε, την συμμετοχή 11 χωρών ε, στο σύστημα, τώρα είναι 20 χώρες ε, και τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια καλή ανταλλαγή πληροφοριών για τα συστήματα επιθεώρησης εργασίας και για τις μεθοδολογίες που ακολουθούνται. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριο Σάγγελ. ευχαριστώ πρόεδρο. Μας δίνετε πέντε λεπτά. Δεν ξέρω, αναερώτηση συνολικά. Προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Er Δεν ξέρω θα αν η ε, συνάδελφό σα με κατάλαβε σωστά. Εγώ είπα ότι υπάρχουν κάποιε χώρε που έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες για τους επιθεωρητές τους, οι οποίες λένε ότι κάνουν τους ελέγχους, δίνουν ε, μια συμβουλή και επιβάλλουν και κυρώσεις σε περίπτωση που χρειάζεται. Νομίζω ότι οι επιθεωρητές εργασίας είναι πάντα εταίροι των εταιριών. Αν κάποιος πει ότι κάτι δεν είναι σωστό, τότε θα πρέπει να του πει και πώς να κάνει το σωστό. Ε, πρέπει να του πει κάποιο ότι ε, ναι, χάλασε το αυτοκίνητο, αλλά το, πρέπει να του πει και πώ το φτιάξει. Η διαπίστωση δεν αρκεί. Αυτό που βλέπουμε συχνά στου ελέγχου, στι επιθεωρήσει, ε, είναι ότι αυτό δεν είναι σωστό, δεν ξέρω τι θα κάνει βρε μια λύση, αν μπορεί να σε βοηθήσει κάποιο, δεν ξέρω. Αυτό συνήθω συμβαίνει. Θα πρέπει να υπάρξει πιο θετική προσέγγιση από την πλευρά των επιθεωρητών να είναι δηλαδή πιο έτοιμοι να δώσουν ε, βοήθεια ε, σε αυτόν που ελέγχουν στις εταιρείε. Αλλά δεν, ε, δεν λέω ότι θα, κάνει, θα πρέπει να κάνουν τη δουλειά της εταιρεία. Όχι, η εταιρεία θα κάνει τη δουλειά της, αλλά χρειάζεται και κάποιος που θα τους βοηθήσει να διορθώσουν το λάθος τους. Κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Euh, Εσείς ε, αναφερθήκατε για το θέμα των ε, κοινωνικών εισφορών ε, και πολλές φορές όταν μιλάμε για μεγάλες επιθεωρήσεις βλέπουμε ότι γίνεται σε συνεργασία με την επιθεώρηση εργασίας αλλά μπορεί να συμμετέχουν και αστυνομικές αρχές ή τελωνιακές αρχές. Πράγματι λοιπόν εκεί Υπάρχει μια συνεργασία. Με συγχωρείτε, δεν το συνηθίζω, αλλά θα σας διακόψω. Γιατί ε, εμείς πήγαμε σε αυτό το εργοτάξιο με τη συνάδελφο και εκεί έγιναν πάρα πολλά θανατηφόρα τυχήματα για να δημοσιευτεί το όλο ζήτημα και μάλιστα αυτό έγινε μέσω μιας αγωνίστριας που κινητοποιήθηκε για να υποστηρίξει τους Πολωνούς εργάτες και ξέρετε απ' έξω όλο αυτό το φάκελο για να τα λέμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, επί, ότι θεωρητικά επί του χαρτού μπορεί να είναι, επί χάρτου μπορεί να είναι καλά τα πράγματα και μπορεί να υπάρχει μια συμφωνία, να γίνονται ε, κάποιες επιθεωρήσεις εργασίας ε, ε, όμως στην πράξη είναι διαφορετικά και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ συχνά είμαστε υπέρ των μεγάλων υπεδομών και των μεγάλων έργων, όμως ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, καλούνται ε, άνθρωποι να δουλέψουν προσωρινά σε αυτά τα έργα και μάλιστα με συμβάσεις ε, οι οποίες δεν καλύπτουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Με συγχωρείτε που σας διέκοψα. Εγώ πιστεύω ότι σε εθνικό επίπεδο λειτουργεί το σύστημα και θα σας πω που εμείς βλέπουμε ένα μεγάλο πρόβλημα και αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα το απόγευμα στη σχέση, ε, στη συνεργασία μεταξύ των διάφορων κρατών. Αν δηλαδή εσείς αναφέρεστε σε πολλούς εργαζομένους, είναι αλήθεια ότι η κοινωνική ασφάλιση μιας χώρας δεν γνωρίζει ποιες συνθήκες εργασίας επικρατούν αλλού. Και αν δούμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, ναι, υπάρχει το σλί, καλά έχουμε στο επίπεδο του ΣΛΙΚ τους διευθυντές των διάφορων επιθεωρήσεων που συνεργάζονται, αλλά στην πράξη υπάρχει πολύ μεγάλη συνεργασία. Ε, δεν υπάρχει συνεργασία γιατί οι άνθρωποι δεν γνωρίζονται, δεν υπάρχει ένα σύστημα πληροφορικής. Έτσι λοιπόν πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Και όταν μιλάμε για την απόσπαση των εργαζομένων, μιλάμε πολύ συχνά για ανοιχτού ή κλειστού καταλόγου. Ξέρετε τα προβλήματα αυτά. Εγώ θα έλεγα ότι αν υπήρχε ένα σύστημα που με κάποιο τρόπο όπου με κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα για τους εργαζόμενους στη χώρα προέλευσής τους, αυτό θα διευκόλυνε πολύ και τις επιθεωρήσεις εργασίας και ε, το έργο της κοινωνικής ασφάλισης. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι σε, εθνικό επίπεδο ε, λειτουργεί καλά το σύστημα εκτός ε, από εκεί που υπάρχουν επιθεωρήσεις μεταξύ των διάφορων περιφερειών, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πρόβλημα. Ich sehe da als einziges Mittel ε, Αυτό λοιπόν νομίζω ότι είναι το μοναδικό εργαλείο που έχουμε για να γίνονται πολλοί έλεγχοι σε μικρά εργοτάξια. Και πάλι έχουμε το πρόβλημα που υπόθηκε. Είναι σαφές ότι αυτοί οι λίγοι που βρίσκονται και στα, που ασχολούνται και με την κοινωνική ασφάλιση και κάνουν και τους ελέγχους, ε, δεν γίνεται να είναι έξι άνθρωποι οι οποίοι θα προσπαθούν να καλύψουν όλα τα εργοτάξια θα πρέπει και σε εθνικό επίπεδο που μπορεί να λειτουργήσει λίγο καλύτερα αλλά και σε διεθνή επίπεδο να υπάρχει δυνατότητα όταν ένας επιθεωρητής επισκέπτεται ένα μικρό εργοτάξιο να έχει τη δυνατότητα να ζητήσει βοήθεια και από το εξωτερικό ή από, την, από άλλη χώρα για να, δουν, ε, για να δει δηλαδή αν αυτός ο εργαζόμενος είναι δηλωμένο, αν όλα βαίνουν καλώ, αν τηρούνται οι προποθέσει κτλ. Εκπαίδευση, αρμοδιότητε που είπα για τους ε, επιθεωρητές τώρα. Ε, δεν ξέρω αν σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να πούμε ότι αυτές θα πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες και αυτή θα πρέπει να είναι η εκπαίδευση. Απλώς λέω ότι στις, σε διάφορες επιθεωρήσεις λείπουν οι άνθρωποι που χρειάζονται για να μπορούν να δώσουν τις σωστές συμβουλές, να κάνουν αποτελεσματικούς ελέγχους. Αυτές είναι, αυτή η εκπαίδευση υπάρχει, δίδεται. Ε, αλλά απλώς δεν υπάρχουν οι εκπαιδευμένοι άνθρωποι σε όλους τους ελέγχους. Αυτό είπα. Ε, <clears throat> θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ähm, λοιπόν, υπήρξαν κάποια ερωτήματα. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Αν αξίζει τον κόπο να επικεντρωθούμε στις ε, υψηλού κινδύνου ε, εταιρείε. Ε, δεν είναι μικρός ο κίνδυνος ωστόσο να ορίσουμε αυτές τις εταιρείε. Να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Στην Βόρεια Γερμανία δίδεται μια σύμβαση σε μια εταιρεία. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν κάποιες εργασίες στην πρώτη σύμβαση που δίνεται στην εταιρεία, στον εργολάβο, αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρξουν δύο γερανοί και άλλα δύο μηχανήματα για να γίνει η δουλειά. Ο... Δίνεται λοιπόν στον υπεργολάβο, ο οποίος όμως έχει μόνο έναν γερανό. Και δίνεται και, και η ίδια σύμβαση σε κάποιον άλλον, ο οποίος έχει τα υπόλοιπα εργαλεία, τα υπόλοιπα οχήματα, συγγνώμη. Υπάρχει όμως, γίνεται ένα τύχημα, υπάρχουν τέσσερις νεκροί, ο ένας είναι εργαζόμενος παράνομα, Νομίζω ότι αυτό είναι ένα αρκετά σύνηθες φαινόμενο και παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στην εργασία. Μιλούμε δηλαδή κυρίως για ε, δραστηριότητες που μπορεί όντως να περιέχουν υψηλό κίνδυνο. Η επιθεώρηση εργασίας βεβαίως ενεπλάκη ε, αφού είχε φύγει ο γερανός, αφού είχε γίνει το δυστύχημα, δηλαδή πολύ αργά. Νομίζω ότι ένας ε, τομέας που θα, μπορούσε, όντως, θα να δράσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το θέμα της πιστοποίησης των ε, εμπειρογνωμόνων που θα πρέπει να έχουν όντως ε, την, ε, τις γνώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν κοινέ αρχές, θα υπάρχει, πρέπει να υπάρχει μια κοινή φιλοσοφία στην, στην επιθεώρηση. Γιατί ακριβώς τις, κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται σε σύνορα είναι πολύ διαφορετικές οι πρακτικές. Ίσως να πρέπει λοιπόν εδώ να προωθήσετε τον ε, ευρωπαϊκό συντονισμό. Και ένα τελευταίο σημείο, νομίζω ότι το θέμα αυτό της ε, ε, ψυχικής επιβάρυνσης δεν είναι τόσο νεφελώδες. Ούτε ζητάει την τεράστια εμπειρογνωμοσύνη Μιλούμε για παραδοσιακούς ε, παράγοντες ε, στρεσογόνους, οι πολύ μεγάλες ε, μέρες, ο πολύ φόρτος εργασίας και το θέμα των πληροφοριών ότι έρχεται ο, άνθρωπος σε επαφή με τους, ε, με τους ε, πελάτες του, πρέπει να δώσει τις σωστές πληροφορίες. Ε, δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να φανταστούμε τι σημαίνει ψυχική επιβάρυνση. το θέμα είναι ότι οι, οι διατάξεις που υπάρχουν λίγουν εκεί που ολοκληρώνονται και οι απαιτήσει για για την εργασία. Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει τίποτε άλλο. θα πρέπει να υπάρξει μάλλον ένας α, κανονισμός για το αντιστρες. Τι σημαίνει α, σωστές συνθήκες εργασίας, τι σημαίνει λαθασμένες συνθήκες εργασίας. Το θέμα δεν είναι να εκπαιδεύσουμε και να βγάλουμε ψυχολόγους στην αγορά. Το θέμα είναι να υπάρχουν κάποιες βασικές κατανοητές αρχές οι οποίες θα ορίζουν τι σημαίνει παράβαση του εργασιακού δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτό το κατόρθωμα τέσσερις ομιλίες σε πέντε λεπτά. Ο Τριόμφ. Θα απαντήσω στο ερώτημα που μου τέθηκε για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιθεώρησης της εργασίας. Όντως αυτό είχα θέσει ως τελευταίο θέμα κι εγώ. Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτον, το θέμα δεν είναι να φανταστούμε ότι αύριο ένας μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός θα υποκαταστήσει τους εθνικούς. Ενώ όμως ότι σήμερα υπάρχουν προκλήσεις πέρα από κάθε έθνος, διαμεθοριακές, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα υπάρχοντα όργανα και οργανισμούς και γι' αυτό νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε τέσσερα πράγματα. Πρώτον, να ορίσουμε κριτήρια του τι εννοούμε ευρωπαϊκή ενωσιακή επιθεώρηση εργασίας. Το SLIC δεν ανταποκρίνεται. Το SLIC ασχολείται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και κατ' παρά το, ε, πέρα από το ότι έχουν φύγει από αυτό πολλά εθνικά συστήματα, έχει ένα προσανατολισμό που, που δεν αναφέρεται αρκετά στο θέμα των βασικών δικαιωμάτων στην εργασία ή των working conditions. Δεύτερον, Νομίζω ότι χρειαζόμαστε πολύ πιο κοινή εκπαίδευση για αυτό το θέμα. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να υπάρχουν κοινά πανεπιστήμια και να μιλάνε όλοι για τον έρασμο, ενώ για τις επιθεωρήσεις της εργασίας να μην έχει γίνει τίποτα τέτοιο. Εξάλλου, οι νεαρότεροι επιθεωρητές και επιθεωρήτριες ε, θα ήθελαν κάποια τέτοια κοινή εκπαίδευση. Τρίτον, τα εργαλεία, τα κοινά εργαλεία. Καταρχήν, οι επιθεωρητές εργασίας δεν θα μπορέσουν να επηρεάσουν τα κέντρα λήψης αποφάσεων αν δεν υπάρχουν πανενωσιακοί κανόνες για τα θέμα της απόδοσης των ευθυνών. Ξέρω ότι το έχετε συζητήσει το θέμα αυτό με αφορμή άλλο κάτι άλλο αλλά πρέπει να πούμε ότι σήμερα δεν υπάρχει ούτε εθνικά ούτε ενωσιακά κάποια τέτοια σύστημα απόδοση φθηνών. Ενώ αν δεν υπάρξει δεν θα μπορέσουμε να επηρεάσουμε καθόλου τις μεγάλες εταιρείες ούτε και το θέμα της υπεργολαβίας. Και καταλήγω με το τέταρτο. Νομίζω ότι τα συστήματα των θεωρητών πρέπει να εξετάσουν τι ωφελεί τους ασθενέστερους και επιχειρήσεις εργαζόμενους και με αυτό θα μπορέσουμε να προσανατολιστούμε. Δεν ξέρω αν χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σώμα επιθεώρησης αύριο, αλλά πάντως δεν θα λυθούν τα τεράστια προβλήματα μόνο με ανεπαρκέστατα το προσωπικό της λεγόμενης αστυνομίας γυτνίασης. Δεν μπορούμε έτσι να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα που ξεπερνούν το τοπικό επίπεδο, ίσως και λόγω της παγκοσμιοποίησης. Κάτω από πέντε λεπτά. Ε. Ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Ξέρετε ότι η θέση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας ποια είναι για την κοινή ευθύνη. Όταν συζητούσαμε την οδηγία για τις αποσπάσεις, ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία της. Και η θέση μας ήταν η πιο προχωρημένη γιατί ξεπερνούσε και αυτά ακόμα που είχε προβλέψει αρχικά η Κομισιόν Ξέρω ότι θα πολύ συζητηθεί πάλι αυτό το θέμα γιατί και σήμερα μόλις το πρωί ακούστηκε επίκριση του Κοινοβουλίου για τη λήψη αυτής της θέσης. Είναι λοιπόν επίκαιρο το θέμα και δεν αφορά μόνο την επιθεώρηση εργασίας αυστηρά, αλλά έχει και άλλα, συνδέεται και με άλλα. Εξ ονόματος λοιπόν όλων των μελών που δεν είναι όλα παρόντα γιατί έχουν και άλλες ενδυμένες προχρώσεις. Σας ευχαριστώ και τους τέσσερις και είμαι βέβαιο ότι η συγγήτρια θα παραμείνει σε επαφή μαζί σας για να επεξεργαστεί συγκεκριμένα θέματα στην έκθεση πρωτοβουλίας της. 26 και 27 Σεπτεμβρίου η επόμενη συζήτηση. Λίγη σύντομα βέβαια η διορία κατάθεση τροπολογιών, αλλά είναι τη λίγη θητεία σε λίγο. 10 Οκτωβρίου στις 12 λίγη. 5 Νοεμβρίου οι τροπολογίες, οι συμβιβασμοί θα υποβληθούν και συζητηθούν στις 25 Νοεμβρίου και την επομένη θα ψηφίσουμε ε, ώστε να περάσει το θέμα στην Ολομέλεια στη Σύνοδο του Ιανού Αρίου. Τελείωσε αυτό το θέμα της ημερήσιας διάταξης. Πάει. Περνάμε τώρα στο 15 και δίνουμε το λόγο στον Φιλ Μπενιόν για το σχέδιο έκθεσής του για την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων στα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. Πρόκειται για έκθεση όπου η Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή είναι συνδεδεμένη με εισηγητή τον Φαβρίκιο Πέρτο του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση αφορά την οικονομική συμμετοχή των υπαλλήλων Φέρουμε σε αυτό ως EFP και νομίζω την ευκαιρία για το Κοινοβούλιο να υπερασπίσει μια πρόταση που να ενισχύει τις επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη, συμμετοχή των ε, εργαζομένων, οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να ωφελήσει και τις επιχειρήσεις ε, αλλά και τους εργαζομένους αλλά και τους ιδιοκτήτες που πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν για τους εργαζομένους Νομίζω ότι λαμβάνω κάποιο feedback. Όχι, χτυπάει ένα τηλέφωνο. Λοιπόν, για τη συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη αποφάσεων ε, για τη δίκηση των επιχειρήσεων, ε, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία μιας ε, μακρόχρονης σχέσης με την εταιρεία και επίσης μπορεί να υπάρχουν και περαιτέρω κίνητρα για τα κέρδη και ε, οι εργοδότες μπορεί να επενδύσουν περισσότερο στην κατάρτιση και για τις εταιρείε και συγκεκριμένα τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η οικονομική συμμετοχή των εργαζομένων μπορεί να παρέχει ένα πόρο χρηματοδότησης που να οδηγεί στη σταθερότητα και φυσικά να καθιστά πιο ασφαλή τις θέσεις εργασίας. Και παρά τα, θετικά είναι σχετικά μικρή συμμετοχή των εργαζόμενων της επιχειρήσης. δεν υπάρχουν ρυθμιστικά κίνητρα, ούτε σαφείς κατευθυντηρίες γραμμές. Στην έκθεση αυτή προσπαθήσαμε να δώσουμε μια σύντομη εξήγηση για ε, το πώς λειτουργούν ε, κάποια ε, τέτοια σχέδια συμμετοχής. Επίσης αναφέρουμε και πώς μπορεί να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στην εξαγορά των επιχειρήσεων και τα διερευνούμε όλα αυτά. Επίσης θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να δούμε το πώς μπορούμε να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε αυτά τα πλεονεκτήματα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και βλέπουμε ένα ισπανικό παράδειγμα των Σοσιαδάδες Λαοράλες Συγγνώμη και για την προφορά μου, λέει ο μιλητή. Αυτό είναι το καλύτερο παράδειγμα στο συγκεκριμένο τομέα. Ένα από τους στόχους της έκθεση είναι να καλέσει να δημιουργηθεί ένα μη δεσμευτικό πλαίσιο για τι αρχέ που πρέπει να διέπουν αυτά τα συστήματα. Αυτέ οι αρχέ συμπεριλαμβάνουν καταρχήν ότι πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο στόχο. θα πρέπει να συμφωνούν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότε για ε, του στόχου του οικονομική συμμετοχής των εργαζομένων τον Δεύτερον, υπάρχει ανάγκη ευελιξίας για να μπορούν να ενταχθούν διάφορα είδη και μεγέθη επιχειρήσεων και διάφορα στόχοι. Θα πρέπει τρίτον να είναι εκούσιο χαρακτήρα, θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν ε, οι εργοδότες αν θέλουν να εφαρμόσουν τέτοιο σύστημα και οι εργαζόμενοι αν θέλουν να συμμετάσχουν σε τέτοιο σύστημα. Τέταρτον, θα πρέπει ε, να, είναι πρόσθετο ε, αυτό το σύστημα στον μισθό μισθό δεν πρέπει να αντικαθιστά το μισθό ή τα σημαντικά δικαιώματα και τέλος θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή παροχή πληροφοριών, θα πρέπει να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι επαρκώς για τις ευθύνε και για τη δικαιώματά του όταν συμμετέχουν σε ένα τέτοιο σύστημα. Επίσης, οι φορολογικές και δημοσιονομικές πολιτικές είναι πολύ σημαντικές για την ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων, αλλά πιστεύουμε ότι και μία ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν ε, είναι κάτι κατάλληλο και η Επιτροπή ΕΚΟΝ εργάζεται επί του θέματος αυτού και περιμένουμε τη γνωμοδότησή τους. Έχουμε οργανώσει διάφορες συναντήσεις με μέρη που ενδιαφέρονται για την έκθεση αυτή και ελπίζουν να μας δώσουν επικοδομητική ανάδραση. Σήμερα αυτή η έκθεση προσπαθεί να παρουσιάσει το δυνατό πιο συγκεκριμένες προτάσεις για να συνεισφέρει στην άνοδο τέτοιων ε, συστημάτων οικονομικής συμμετοχής των εργαζομένων και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους από εδώ και πέρα. Άγνερ και στη συνέχεια Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μπενιόν για την δουλειά που έκανε. Είναι όντως πολύ επικοδομητικός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το θέμα. Για την συμμετοχή λοιπόν των εργαζομένων, ε, νομίζω ότι είναι ένα πολύ εξειδικευμένο θέμα. Υπάρχουν τόσα πολλά διαφορετικά μοντέλα που μπορεί να λειτουργούν καλά σε κάποια εταιρεία, σε κάποια άλλη μπορεί να μην λειτουργούν. Θα ήθελα να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολύ ε, κατακριματισμένες πρακτικές ε, η έκθεση όμως είναι μια πολύ καλή βάση για να μπορέσουμε να σχολιάσουμε το θέμα αυτό. Ε, για την πρόταση που κάνει τώρα ο κύριος ε, Μπενιόν για την προαιρετική δημιουργία αυτού του 21ου καθεστώτος ας πούμε συστήματος. Είναι μια πολύ καλή ιδέα αυτή με βάση λοιπόν και την πρακτική εμπειρία που έχουμε θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε αλλά ακόμα νομίζω ότι δεν είναι τόσο όριμα τα πράγματα. Τώρα για το ποια θα είναι η καταλληλότερη λύση, ε, ίσως μια προτροπή του Συμβουλίου προς τα κρατη σε αυτό το στάδιο να τους προτείνει κάποιες, κάποιους τρόπους αντιμετώπισης, ίσως θα μπορούσε να τους δώσει και κάποια παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για να συνδυαστούν λίγο όλες αυτές οι διαφορετικές πρακτικές που υπάρχουν. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουμε διαφήμιση για τις δυνατότητες που υπάρχουν συμμετοχή των εργαζομένων. Ή θα πρέπει να υπάρξει ξέρω εγώ, μια γραμμή του προπολογισμού που θα δώσει η Κομισιόν ή μια εκστρατεία. Θα πρέπει να σκεφτούμε. τώρα, εκεί που δεν υπάρχει συμμετοχή των ε, εργαζομένων, ίσως ας πούμε στις ε, χώρες της Κεντρικής ή Ανατολικής Ευρώπης, εκεί που δεν υπάρχει πώς θα μπορούσε να προωθηθεί. Ο κύριος Μπενιόν ε, μίλησε και για τα φορολογικά θέματα. Αυτό βεβαίως είναι θέμα ουσίας. Δεν χρειάζεται να το λέμε. θέλουμε ευρωπαϊκά να το δούμε το θέμα αυτό. Και αν δεν υπάρξει ε, έτσι, συνεννόηση μεταξύ των κρατών μελών, προφανώς και το 21 ο σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε δεν θα έχει καμιά επιτυχία. Και τα πιο σημαντικά σημεία ε, είναι η ε, ανεξαρτησία, ε, προσαρμογή στις κατατόπους απαιτήσεις και επίσης θα πρέπει να ε, θέλουν και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν. Αυτό βεβαίως θα πρέπει να γίνει και μέσω συμβουλών και μέσω διαβουλεύσεων. Ούτως ή άλλως και ο κύριος Μπενιόν το αναφέρει στην εκθεσή του. Ε, εγώ θα ήθελα εδώ απλώς να μιλήσω για την παράγραφο 12 συγκεκριμένα, όπου μιλάει για μια αλλαγή των συνδικάτων προς, την, ε, προς αυτή την κατεύθυνση έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, ε, νομίζω ότι έχει θετική ε, πρόθεση με αυτό που λέει ο κύριος Μπενιόν, αλλά ίσως εδώ να πρέπει να αλλάξουμε λίγο την διατύπωση. Ε, μπορεί να μην δίνουμε το σωστό μήνυμα. Ίσως δηλαδή να δίνουμε την εντύπωση ότι βασιζόμαστε πάνω σε αυτές τις διαφορές που υπάρχουν ένα κράτος μέλος για να μην προωθήσουμε ε, τη συμμετοχή των ε, εργαζομένων. Ε, πέραν αυτού, ε, εγώ χαίρομαι για τις ε, συζητήσεις που θα κάνουμε. Ήδη έχει γίνει πολύ καλή, πολύ επικοδομητική δουλειά. Έχουμε κάνει πολύ καλή ανταλλαγή απόψε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είμαι σκιώδης ε, του ΕΛΚ. Απλά θα ήθελα να κάνω κάποια προσωπικά σχόλια. Ελπίζουμε, ελπίζω να διατηρήσουμε την, ε, τον ακούσιο χαρακτήρα της έκθεσης αυτής και να γίνει σεβαστή και η αρχή της επικουρικότητας, ε, την επικουρικότητα των κρατών μελών, όπως και την επικουρικότητα των εταιριών. Είμαι κάπως σκεπτική για το σημείο 7 και 8 δηλαδή για ένα μοντέλο σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Καθώ ακούσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά είδη μοντέλων. ίσω η ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών ε, να λειτουργήσει καλύτερα εδώ. Και στο σημείο 11 ε, υπάρχουν αυτά τα αλφαβήτα γάμα και όπω σα είπα θα πρέπει εδώ να τονιστεί ο εθελοντικό και μη υποχρεωτικό χαρακτήρα. Ευχαριστούμε. Κύριε Σεργέν για την, Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια για τη δουλειά της που συμφωνεί με αυτά που συζητούμε και εμείς στη Γενική Διεύθυνση Αγορών για τη συμμετοχή των εργαζομένων. Το τελευταίο νέο είναι ότι άρχισε ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα άρχισε την επόμενη Δευτέρα που ακολουθεί η εκθεσή σας. Ελπίζουμε δηλαδή να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Πρώτον ένα mapping όλων των διαφορών μεταξύ χωρών που αναφέρατε και που να εξηγήσει, αν εξηγεί, τις διαφορές μεταξύ τους και επίσης το 21ο καθεστώς ή η χρησιμοποίηση των building block μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο. Θα δούμε τι θα μας δείξει η ανάλυση και μέσα στον Ιανουάριο θα γίνουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε για αυτές τις αποσαφηνήσεις. Τώρα ξανά ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ. Θα σχολιάσω αυτά που ακούστηκαν. Η κυρία Ρέγνερ μίλησε για μια καμπάνια πληροφόρησης για να διαδοθεί η ιδέα αυτή. Πολύ χρήσιμο νομίζω θα ήταν να το εξετάσουμε. Δεν χρειάζεται να είναι απλώς πληροφόρηση, αλλά θα μπορούσαν και οι ενδιαφερόμενοι ίδιοι να συμμετάσχουν place. Um, on the 19th, uh, uh, Έχουν ήδη γίνει προταθεί 29 τέτοια προγράμματα και ακούστηκαν ήδη πολλές αμφιβολίες και πρέπει να ομολογήσω και εγώ ότι δεν είμαι βέβαιος για το κατά πόσον μπορεί, είναι εφαρμόσιμο. Υπάρχουν εταιρείες που ξεπερνούν τα εθνικά σύνορα, είναι σαν πανενωσιακές εταιρείες και είναι δύσκολο όταν είναι τόσο διαδεδομένη ή ευρεία η εργατική δύναμη, το εργατικό δυναμικό είναι δύσκολο να νομοθετήσουμε γι' αυτό γενικότερα. Αλλά θα δούμε αν είναι δυνατόν ή όχι. Θα ήθελα, αλλά αναγνωρίζω από τώρα ότι θα υπάρξουν πρακτικές δυσκολίες. Τώρα εδώ μάλλον κάνω μια υπόθεση ότι γιατί στο Ηνωμένο Βασίλειο εμείς αυτά τα βλέπουμε πιο θετικά ίσως στα συνδικάτα τουλάχιστον. Πάντοτε ήταν έτσι. Ίσως να αλλάξω τη διατύπωσή μου εκεί που τα λέω αυτά, αλλά είναι αλήθεια. Ότι τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη αποδοχή της ιδέας αυτής και ακούγονται ιδέες για συνδυασμένη διαχείριση εργαζομένων εργοδοτών ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι εταιρείες δεν βρίσκουν διάδοχο και όπου οι εργαζόμενοι προτιμούν να συνεχίσουν τη δραστηριότητα της εταιρείας παρά να εξαγοραστούν από κάποια άλλη εταιρεία και να εγκατασταθούν αλλού. Σε αυτό το τομέα νομίζω μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Αυτά γίνονται όλο και συχνότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και εξετάζοντας τις βέλτιστες πρακτικές μπορούμε να πάρουμε και άλλα παραδείγματα. Μάλιστα, καλή βάση όλα αυτά για την περαιτέρω συζήτηση. Η ωραία κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 10 Οκτωβρίου το μεσημέρι. Θα εξετάσουμε τις τροπολογίες στις 5 Νοεμβρίου συμβιβαστικές 25 και η ψηφοφορία στις 5 Δεκεμβρίου για την Ολομέλεια του Ιανουαρίου ή του Φεβρουαρίου. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 16, στα σημεία 16 και 17 και άρα θα δώσω το λόγο στον Φρεντερίκο Ντάρντεν που θα γνωμοδοτήσει για την Επιτροπή Μεταφορών στα δύο κείμενα δηλαδή της λεγόμενης σιδηροδρομικής δέσμης, η πρώτη τροποποίηση του κανονισμού ειδικά με το άνοιγμα της αγοράς εγχώριων επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών 1370 κάθετος 2007 και το δεύτερο κείμενο είναι η τροπή της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροπο, τροποποιεί την οδηγία 2012-34 της 21 η Νοεμβρίου 2012 για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου όσον αφορά το άνοιγμα της αγοράς εσωτερικών σιδηροδρομικών επιβατικών μεταφορών και τη διακυβέρνηση της σιδηροδρομικής υπαδομής. Ορίστε κύριε εισηγητά μου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα κάνω μια καθολική παρουσίαση για το πνεύμα αυτών των δύο με δύο λόγια. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω το και μάλλον ε, το εκφράσετε, το διαβάσατε και στην συντομητιολόγηση ότι δεν είμαι πεπισμένος για την αναγκαιότητα περαιτέρω απελευθέρωσης ε, του συνδρομικού τομέα μέσω αυτού του τέταρτου συνδρομικού πακέτου. Ακόμη ε, δεν ε, έχουμε σημαντική οπισθοχώρηση σε σχέση με το τρίτο πακέτο και ε, επομένως δεν είμαστε πεπισμένοι από αυτή την ευκαιρία. Αλλά ευθέντως αυτού είχαμε δύο δυνατότητες αυτές ε, δύο δυνατότητες, ε, είτε να έχουμε μια γνωμοδότηση και να προτείνουμε την απόρριψη αυτού του τέταρτου πακέτου, της τέταρτης μέτρων, ή να είμαστε πιο επικοδομητικοί στην προσέγγισή μας. Επιλέξαμε να καταθέσουμε μια γνωμοδότηση με διάφορες προτάσεις. Ε, πράγματι, τελικά βλέπουμε ότι είναι πολύ μικρή η δυνατότητα, η πιθανότητα να απορριφθεί το κείμενο στην Επιτροπή Μεταφορών. Γι' αυτό και εγώ επέλεξα τη λογική αυτή που μου φαίνεται πλέον κατάλληλη. Έτσι λοιπόν στα πλαίσια αυτής της λογική θέλαμε να παρουσιάσουμε ένα κείμενο που να τροποποιεί την πρόταση της Κομισιόν σε ό,τι αφορά κάποια στοιχεία που θα σας τα παρουσιάσω Κατ' Καταρχήν μεγάλη προστασία των επιβατών. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο και αν δεν προέρχεται από τη δική μα Επιτροπή δεν ξέρω από πού θα προέρθει. Έτσι λοιπόν ε, μεγάλη προστασία των εργαζομένων για το είναι μετάβαση ε, των εργαζομένων από τις ιστορικές επιχειρήσεις στις νέες επιχειρήσεις με τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προστατεύσουμε τις συνθήκες εργασίας όποιο και αν είναι το καθεστώς αυτών των εργαζομένων. Επίσης, μεγαλύτερη ελευθερία στην Εθνική Ρυθμιστική Αρχή για να επιλέξει την άμεση ανάθεση παρά τους διαγωνισμούς. Και έχουμε μια τροποποίηση σε σχέση με το νότο και σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς απόλυτης ελευθερίας. Αυτό είναι μια δεύτερη θεματική. Τρίτη θεματική, μεγαλύτερη ελευθερία σύνδεσης ε, μεταξύ των στοιχείων του χαρτοφυλακίου, δηλαδή να μειώσουμε τις υποχρεώσεις ε, ε, περιορισμού σε άξονες προτείνεται η μεταρρύθμιση από την Κομισιόν και επίσης να έχουμε και μία και μεγαλύτερο χρόνο για την εφαρμογή αυτού του τέταρτου πακέτου. Νομίζω ότι στις 25 του μήνα είναι προθεσμία κατάθεση τροπολογιών και βέβαια δεν αποκλείω να καταθέσω και άλλες τροπολογίες για να ενισχύσω αυτές τις ε, πτυχές που σας ανέφερα, αλλά φυσικά περιμένω και τα σχόλια των συναδέλφων για να δούμε αν θέλουν να συζητήσουμε κάτι περισσότερο εις βάθος. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ η κυρία Σπακ και κατόπιν η κυρία Στέτερ. Συγγνώμη κύριε Σπακ, ευχαριστώ. Για το τέταρτο πακέτο για τους ε, σιδηροδρόμους εκτιμώ τις ε, εξηγήσεις του εισηγητού ε, και εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό και οι προτάσεις της Κομισιόν Θεωρώ ότι θα, θα δημιουργούσαν πρόβλημα αν περάσουν όσα έχουν και για τους απασχολούμενους στον τομέα και για τους επιβάτες. Είναι καλό λοιπόν που και η Επιτροπή Τραν αλλά και η Επιτροπή Απασχόλησης θα υποβάλουν τις σχετικές τροπολογίες. Για τις προτάσεις πρέπει να πω ότι η στοχοθέτηση, η κατεύθυνση δηλαδή είναι σωστή ε, για αυτή την απελευθέρωση των εθνικών δικτύων ε, ε, θα πρέπει να αποφευθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ και αυτό ισχύει και για τις δύο προτάσεις και τις δύο εκθέσεις. Ένα βασικό σημείο σε τούτο τον κανονισμό είναι το θέμα της ελεύθερης επιλογής. Γιατί μιλούμε και για το θέμα των άμεσων αναθέσεων και ο Φεντερίκ Νομίζω ότι πολύ σωστά το λέει, το είπε και στην αρχή. Υπάρχει και η πρωτοβουλία α, να υπάρξει ε, απόρριψη, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσει πολύ εύκολα αυτό. Αλλά στο μέλλον θα πρέπει να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν ελεύθερα εάν θέλουν να συνεχίσουν με τις άμεσες αναθέσεις ή αν θέλουν να κάνουν διαγωνισμούς. Και στην τροπολογία 5, για αυτή την αμοιβαιότητα, όπου μιλούμε και για τις τρίτες χώρες και που πρέπει να πληρούν και αυτές τις ίδιες προϋποθέσεις με μας, ε, νομίζω ότι αυτό δεν πάει πολύ μακριά. Ε, Εντό της Ένωσης μιλούμε για κοινωνικό dumping, όπου οι μεγάλες εταιρείε μεθυγατρικές ε, κάνουν διάφορες μεταφορές και παρόλα αυτά δεν τηρούν τις προϋποθέσεις οι οποίες υπάρχουν, δίνουν τις συμβάσεις κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την τροπολογία και στις, ε, στις και όχι μόνο στις μητρικές εταιρείες. Επίσης οι υπεργολάβοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν εδώ. Νομίζω ότι είναι καλό αυτό, στην τροπολογία 22 το λέει. Ίσως ο εισηγητής θα μπορούσε να μας δώσει πιο συγκεκριμένες συστάσεις ή θα μπορούσαμε ίσως ε, να ελουδίσουμε λίγο το κείμενο, δεν είναι απόλυτα σαφές για μένα. Μετά μιλούμε για τη διακυβέρνηση. Η άνοιξη, το άνοιγμα της αγοράς νομίζω ότι δεν πρέπει να σημαίνει ενιαίο ε, μοντέλο για όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, διαφορετικά μοντέλα για τα μικρά κράτη-μέλη και τα μεγάλα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε τα μεν με τα δε υπάρχει, υπάρχει απόλυτη απελευθέρωση, υπάρχουν τα holdings, υπάρχουν διάφορα συστήματα λοιπόν, εφόσον, ε, τηρούνται οι εφόσον πληρούνται οι προποθέσει για την αποφυγή ε, του dumping. Αλλά τώρα ενιαίο μοντέλο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Επίση, ο κοινωνικό διάλογο ε, είναι πάρα πολύ σωστό και η οπτική γωνία από την οποία το βλέπει ο Φρεντερίκ είναι πολύ σωστή. και για το προσωπικό αυτό που αναφέρει στην έκθεσή του είναι σημαντικά, και αυτός επίσης και για τις ε, δεσμολογικές ε, συμβάσεις ε, και αυτό που λέει επίσης είναι άξιο λόγου. Υπάρχουν λοιπόν πολλά κοινά σημεία πάνω στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, ο Φίλιππος Ντεμπάκερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή για την παρουσίαση και τις προτάσεις του. Δεν θα σας εκπλήξει το γεγονός ότι όπως ξέρετε εγώ έχω μια πολύ στεναρή θέση για το θέμα αυτό γιατί όλοι φαίνεται να συμφωνούν ότι πρέπει να κινηθούμε με μια κατεύθυνση που, με την οποία εγώ διαφωνώ. Θα εξηγήσω. Θα τα εξηγήσω μάλλον στις τροπολογίες που θα καταθέσω. Οι σιδηρόδρομοι έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια λόγω του ανταγωνισμού με άλλες μορφές μεταφορών. Και ο λόγος για μένα είναι φανερός. Εάν οι σιδηρόδρομοι δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί και ευέλικτοι με τους επιβάτες τους, τότε θα χάσουν βέβαια ελκυστικότητα. Και άρα αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορέσουμε να προωθήσουμε, να βελτιστοποιήσουμε τη χρήση των σιδηροδρόμων. Δεύτερον, οι προτινόμενες τροπολογίες από τον εισηγητή, μερικές τουλάχιστον, βασίζονται μάλλον σε ιδεολογία παρά στα γεγονότα. Ένα παράδειγμα, μιλάει για τον κίνδυνο του κοινωνικού ντάμπινγκ, της απώλειας θέσεων εργασίας, απολύσεων, λόγω των αλλαγών αυτών. Θα ήθελα να του υποδείξω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία είναι οι μόνες χώρες που προσέλαβαν περισσότερους στους σιδηροδρόμους από ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες που απολύουν. Αυτό αποδεικνύει ότι η απελευθέρωση και το άνοιγμα της αγοράς δεν σημαίνει αναγκαστικά απώλεια θέσεων εργασίας και κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό φαίνεται και από τους αριθμούς, από τους μισθούς δηλαδή των σιδηροδρομικών. Ο μέσος μισθός είναι ψηλότερος στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία από ό,τι στη Γερμανία. Ακόμη μια φορά λοιπόν δεν συνδέονται τα δύο θέματα απελευθέρωση με ανεργία. Φέρε την ασφάλεια τα ίδια. Αν δούμε τα τελευταία δέκα χρόνια σε ορισμένες χώρες που άνοιξαν τα σιδηροδρομικά του συστήματα είναι σήμερα οι καλύτεροι μαθητές της τάξης ως προς την ασφάλεια. Για τη διαχείριση επίσης διαφωνώ. Υπάρχει διαφορά μεταξύ της δουλειάς που πρέπει να κάνει ένας λειτουργικός διαχειριστής με έναν διαχειριστή του υλικού. Είναι λογικό να διαχωριστούν οι δύο δραστηριότητες λοιπόν. Πώς, με τα συμβόλαια, τη συνεργασία, οτιδήποτε. αλλά νομίζω ότι ο διαχωρισμός των δύο εργασιών είναι ουσιώδης. Όπως γίνεται και στη χώρα του εισηγητή. Αυτά είναι οι σκέψεις μου. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε επικοδομητικό ρόλο στη συζήτηση αυτή, αν και θα διαφωνήσουμε, αλλά θα είμαστε επικοδομητικοί στις προσπάθειές μας να καταλήξουμε σε μία σωστή γνωμοδότηση. Εμείς θέλουμε άνοιγμα της αγοράς για ασφαλέστερους σιδηροδρόμους και καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και επιβατησών. Ευχαριστώ. Η Ελίζα Μπετστρότερ. Ευχαριστώ. Και εγώ είμαι επικριτική απέναντι στην πρόταση Κομισιόν, γιατί βλέπω ότι δεν είναι σαφές γιατί έρχεται τώρα αυτή η πρόταση, γιατί πρέπει να γίνουν τώρα αυτά τα πράγματα. Ακόμη δεν έχουμε εφαρμόσει την οδηγία, ακόμη δεν έχουμε συλλέξει εμπειρίες από την εφαρμογή της οδηγίας. Έχω την εντύπωση ότι ο λόγος για τον οποίο γίνεται τώρα αυτό είναι μια στοχευμένη πίεση για απελευθέρωση. Και δεν νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει να βελτιωθεί η ποιότητα. Η ποιότητα θα γίνει καλύτερη εκεί που αξίζει, δηλαδή στα κέντρα. Σε μεγάλες όμως απομακρυσμένες περιοχές δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει. Με μονομένες ε, λύσεις είναι αυτές που θα βοηθήσουν ε, να, διατηρηθεί, να, διατηρηθούν οι μεταφορές σε αυτές τις περιοχές. Η δική μας η αρμοδιότητα είναι να ασχοληθούμε με το θέμα της προστασίας του ε, εργαζόμενου. Και ως προς αυτό στην πρόταση Κομισιόν δεν υπάρχει τίποτε. Μάλλον θα πρέπει λοιπόν να προσθέσουμε σημεία ε, επιπλέον στην ε, πρόταση έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις για τους εργαζόμενους. Υποστηρίζω λοιπόν την πρόταση του εισηγητή να διατηρήσουμε για ακόμη περισσότερο την ε, μεταβατική περίοδο. Πρέπει επίσης να ε, έχουμε ολοκληρωμένες λύσεις, το είπε και ο συνάδελφος Μπαχ, πιο επικριτικά βλέπω τον άλλο φάκελο ωστόσο, το άνοιγμα της αγοράς για τις ε, μεταφορές, για τις μετακινήσεις. Ε, εκεί, ε, μάλλον το θέμα αυτό το έχει συζητήσει και ο συγκεκριτής πολύ, το θέμα είναι οι ε, συνέπειες του ήδη υπάρχοντος ανοίγματο της αγοράς, γιατί μιλούμε για πάρα πολύ προσωπικό, το οποίο είναι, δεν είναι εκπαιδευμένο, δεν είναι εξειδικευμένο, σημαίνει αυτό λιγότερη ασφάλεια, σημαίνει αυτό χειρότερη ποιότητα παροχής υπηρεσιών, και βεβαίω υπάρχει ανισορροπία, σαφώ μεγαλύτερη ανισορροπία μεταξύ των αστικών χώρων και της υπαίθρου. Και αυτό βεβαίως αντίκειται και στους στόχου τη Ευρωπαϊκής Ένωση, αντίκειται στους στόχου ε, του κοινωνικού τη ευρωπαϊκή ένωση, και θεωρούμε ότι είναι απολύτως σαφέ, ότι οι μεταφορέ θα πρέπει να δομηθούν με τέτοιο τρόπο και αυτό είναι όντω στόχο που θέλουμε να υπάρξει, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας ανεξάρτητα από το κοινωνικό του στάτους να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το είδος μεταφορών και να μην ε, ορίζεται αυτό από την ε, τιμή που θα καθοριστεί. Δεν πρέπει να είναι ε, είδος πολυτελείας οι μεταφορές, προφανώς ο καθένας, ανεξάρτητα που μένει και πόσα χρήματα έχει στην τσέπη του, θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα μεταφοράς. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν στην έκθεση. Εγώ ε, τρόμαξα όταν είδα το σχέδιο της ε, πρότασης της Κομισιόν. Η Κομισιόν έκανε μια πολύ διαφορετική συζήτηση σε ό,τι αφορά το πρώτο άνοιγμα που κάναμε τη συζήτηση εδώ και είχαμε πει ότι πρέπει να φροντίσουμε και τότε την ε, πρόσβαση σε όλους ανεξάρτητα της κοινωνικής τους ε, τάξης. Και αυτό δεν είναι ληφθή υπόψη. Ε, έγινε πολύ μακρά συζήτηση, το Κοινοβούλιο έκανε πολύ συγκεκριμένε προτάσει και πήρε πολύ συγκεκριμένε αποφάσει και η Κομισιόν έρχεται τώρα, τα βάζει όλα στην άκρη και υποβάλλει μια δική τη πρόταση. Ε, χαίρομαι που ο συνάδελφο ε, Μπαχ είναι σκιώδη ηγητή σε αυτό, είναι και στην Επιτροπή Μεταφορών, ξέρει την συζήτηση που γίνεται και εκεί, οπότε μπορούμε από κοινού να το σκεφτούμε, να συζητήσουμε, να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε σε αυτό το φάκελο αυτά που θέλουμε. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε με, με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουμε με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπενιόν. Αλλά να δώσω και το λόγο στην Κομισιόν, όχι, ο κύριος Μπενιόν. Θα ξεκινούσα με τα αριθμητικά στοιχεία που παρουσίασε ο κύριος Δεμπάκερ για τις χώρες που έχουν προβεί στην απελευθέρωση. Εγώ ζω σε μία από αυτές τις χώρες, όπου διπλασιάσαμε τον αριθμό των επιβατών στους σιδηροδρόμους από τις αρχές ε, του 2000 ε, ε, και από το 99 μέχρι σήμερα, σε 14 χρόνια, διπλασιάσαμε τον αριθμό των επιβατών και φυσικά υπήρξε και αύξηση των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους και κατά μέσο όρο έχουν βελτιωθεί οι μισθολογικέ του συνθήκες σε σχέση με το υπόλοιπο εργατικό δυναμικό. Έτσι λοιπόν οι φόβοι που εκφράστηκαν, γιατί έτσι του θεωρώ, είναι αβάσιμοι. Και είχαμε και την ίδια συζήτηση το 1996 όταν συζητούσαμε αυτή τη διαδικασία για τα πρώτα τρία-τέσσερα χρόνια. Ε, τα είχαμε ε, μπερδέψει για τα όλα ζητήματα, αλλά τελικά αυτό που προτείνει τώρα η Κομισιόν δεν είναι αυτό που προσπάθησε να γίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1996, είναι πως ε, διορθώσαμε την κατάσταση υπό το φως της εμπειρίας που είχαμε. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν προτείνει ένα σύστημα πολύ παρόμοιο με το σύστημα που απολαμβάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο που είδαμε μεγάλη αύξηση του αριθμού των επιβατών, πολύ μεγάλη αύξηση των αριθμών των εργαζομένων στους σιδηροδρόμους και ε, εκεί που ήμασταν από τους ε, από αυτούς που είχαν τη χειρότερη ποιότητα στην αξιοπιστία του συστήματος, τώρα είμαστε από τους καλύτερους. Και ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά και θα σας παρουσιάσω μια προσωπική εμπειρία. Αυτή η προσέγγιση λειτουργεί για την υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας, ε, όπως και για την ανοιχτή πρόσβαση. Εγώ στο δικό μου σταθμό υπάρχουν δύο γραμμές, μία περνάει προς το Λονδίνο και άλλη προς το Μπέρμπιχαν. Πριν από την ιδιωτικοποίηση είχαμε πέντε τρένα την ημέρα μπορούσα να, με τα οποία μπορούσα να φτάσω στο Λονδίνο. Τα δύο έπρεπε να σταματήσουν να πάρω λεωφορείο, ε, χρειαζόμουν δυόμιση ώρες ε, και ήταν ακριβά. Ξακολουθεί να είναι ακριβό το εισιτήριο βέβαια, αλλά αυτό δεν το έχουμε λύσει ακόμη γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότηση της κυβέρνησης για να υποστηρίξει τις τιμές των εισιτηρίων. Αυτό είναι διαφορετικό θέμα βέβαια. Όμως τώρα για τη γραμμή του Λονδίνου έχουμε μία υπηρεσία τρένο κάθε ώρα και έλεγαν στην αρχή ότι δεν υπήρχε αγορά. Όμως τελικά έχει πάρα πολύ κόσμο και κοστίζει 30 λίρες, ένα στρίο μεταπιστροφής στο Λονδίνο είναι 200 χιλιόμετρα. Δεν νομίζω ότι είναι λοιπόν πολλά 40 ευρώ για 200 χιλιόμετρα και έτσι λοιπόν έχουμε τώρα τόσα πολλά απευθείας ε, τρένα, ενώ στο παρελθόν δεν είχαμε απευθείας τρένα. Και πάλι στην άλλη γραμμή το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε τρένο κάθε μισή ώρα είναι ο υπερ, είναι υπερβολικός αριθμός επιβατών. Νομίζω λοιπόν ότι δεν έχουμε τίποτα να φοβόμαστε γιατί κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία, στην αρχή κάναμε πολλά λάθη, τα διορθώσαμε όμω, αλλά σίγουρα δεν θα με τώρα. Έχουμε ένα πολύ καλύτερο συνομικό σύστημα από ό,τι στο παρελθόν και σε ό,τι αφορά την άμεση ανάθεση, νομίζω ότι το πρόβλημα με την άμεση ανάθεση είναι η έλλειψη εμπιστοσύνη και διαφάνειας γιατί πραγματικά παρεμποδίζονται ε, νέοι φορείς να συμμετέχουν στο σύστημα. Εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες άμεσες αναθέσεις, αλλά χρησιμοποιούνται κυρίως αν χρεοκοπήσει κάποια εταιρεία και πρέπει πολύ γρήγορα να αντικατασταθεί από μια νέα εταιρεία. Αυτά ε, είναι κάποιε χρήσιμε λύσεις, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν σταματά η παροχή υπηρεσιών, δεν σταματούν οι υπηρεσίες. Γενικά είναι καλέ οι προτάσει της Κομισιόν, αν και εμείς από την Επιτροπή Μεταφορών έχουμε υποβάλει πάρα πολλές ε, τροπολογίες για να είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιώσουμε το κείμενο που μας παρουσιάστηκε. Δεν είναι όλα αρνητικά λοιπόν. Υπάρχουν και κάποια καλά για το προσωπικό στα τρένα επειδή είναι επαγγελματίε και στο Ηνωμένο Βασίλειο έτσι του συμπεριφερόμαστε ως επαγγελματίε και οι διοικητέ των τρένων είναι άνθρωποι με πολύ ψηλή κατάρτιση. Το τελευταίο σχόλιο αν ε, διατηρήσουμε ένα κατακαιρματισμένο σύστημα, τότε θα αποτύχουμε εντελώς ε, στο να υπάρχει μετακίνηση του μοντέλου από τις χερσαίες μεταφορές ε, στις συνδρομικές μεταφορές. Από τις οδικές μεταφορές, με συγχωρείτε, στις συνδρομικές μεταφορές. Ο προστατευτισμός σε εθνικό επίπεδο απλώς θα σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει γιατί θα παρουσιάζονται λόγοι κλειστών αγορών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Να δώσω το λόγο στην Κομισιό. Συγγνώμη, κυρία, με συγχωρείτε. Good afternoon. I'd like to thank the... Καλησπέρα σας να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τα δύο σχέδια εκθεσεών του και τα... ευχαριστώ όλους για τα σχόλιά τους. Η Κομισιόν ε, φέλεξε ένα πολύ, ε, μια πολύ ισόρροπη ε, και σταδιακή προσέγγιση για να ανοίξει τις αγορές στο, στις μεταφορές, στον ανταγωνισμό. Ε, θέλουμε να διατηρήσουμε τα ε, πλεονεκτήματα βεβαίω που έχουν τα κράτη-μέλη και τις αρμοδιότητες που έχουν να ορίζουν από μόνα τους ε, κάποιες συνθήκες. Θέλουμε να υπάρξει ισορροπία, θέλουμε να προστατεύσουμε την οικονομική βιωσιμότητα των συμβάσεων δημοσίου τομέα η προτινόμενη εισαγωγή των ε, διαγωνισμών για, τον, ε, για την απόδοση των συμβάσεων θα διευκολύνει τις αρμόδιες αρχές να κάνουν εξοικονόμηση πόρων μέχρι 20-30% και να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρόταση αφήνει περιθώριο λιγμών στα κρατημέλη και στις αρμόδιες αρχές να ορίσουν το σύστημά τους ε, σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών τους. Οι κοινωνικές συνέπειες της πρότασης είναι, σαφές, είναι σαφώς ένα θέμα για, τον, ε, για την Επιτροπή σας και για τον εισηγητή. Η, αν το τέταρτο πακέτο της, ε, της Κομισιόν θα οδηγήσει σε ανεργία ή αν θα μειωθούν οι μισθοί. Το άνοιγμα της αγοράς δεν σημαίνει ανεργία, όπως είπε ο κύριος Δουμπάκερ και ο κύριος Μπανιόν. Η ανεργία στον ε, κλάδο έχει μειωθεί σε όλα τα κρατημέλη σχεδόν. Παρ' όλα αυτά, σε δύο κρατημέλη που έχουν ανοίξει τις αγορές τους στην, ε, στον ε, ανταγωνισμό, οι ε, εργαζόμενοι γίνονται όλο και περισσότεροι. Το άνοιγμα λοιπόν στον ανταγωνισμό μπορεί να δημιουργήσει νέε υπηρεσίε, άρα νέε ε, και πιο εξειδικευμένε θέσει εργασία. Επίση, η πρόταση ε, διευκολύνει περισσότερο, τις, μάλλον απαλύνει τι συνέπειε που υπήρχαν σε σχέση με την προσέγγιση που έχουμε μέχρι τώρα για το άνοιγμα των αγορών. Έχουμε την 34 του 2012 οδηγία που έχει τις ε, σχετικές προτάσεις για την, με τις, μέσω, των προτάσ, μέσω των τροπολογιών 1, 15, 4, 5 και 14. Ε, η Κομισιόν θεωρεί ότι, κάποιες, ε, ότι αν υπάρξουν πολλές τροπολογίες δεν θα βοηθήσει αυτό στην διευκόλυνση των μετακινήσεων και των μεταφορών. Θα πρέπει να υπάρξει για τα κράτη-μέλη ευελιξία θα πρέπει να τονιστεί ο διαχωρισμός και οι σχετικέ απαιτήσει που υπάρχουν και ότι αυτό προτείνεται μόνο για να εξασφαλίσουμε άμεση ίση πρόσβαση σε όλους τους operators στο δίκτυο. Η Κομισιόν προτείνει ευελιξία σε αυτό το είδη των υποδομών, ε, ζητά οικονομική διαφάνεια και, να υπάρξει αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων μέσω των τροπολογιών 11 και, 13 γίνεται αυτό. Θα, δεν θέλουμε να υπάρξει περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά Ήδη υπάρχουν δυνατότητες ε, αποκλειστικών δικαιωμάτων ε, για ε, σχετικές συμβάσεις που πρέπει όμως να είναι σαφώς καθορισμένες και αναλογικές. Το σχέδιο έκθεσης για τον κανονισμό PSO περιλαμβάνει κάποιες τροπολογίες που βελτιώνουν την, κατάσταση όπως η 27 και η 25. Επίση, υπάρχουν κάποιες σχέδια τροπολογιών που η Κομισιόν δεν μπορεί να υποστηρίξει. Σε ό,τι αφορά την απόδοση των συμβάσεων PSO, ο εισηγητή λέει να διατηρηθεί η επιλογή μεταξύ άμεση ανάθεση και ανάθεση μέσω διαγωνισμού η Κομισιόν θεωρεί ότι οι διαγωνισμοί θα πρέπει να αποτελέσουν τον κανόνα. Όπω είπαμε πιο πριν, η εμπειρία δείχνει ότι η ανάθεση συμβάσεων μετά από διαγωνισμού οδηγεί σε κέρδη 20-30%. Ε, πέραν αυτού, η αποτελεσματικότητα τη αγορά σιδηροδρόμων θα βελτιωθεί μόνο αν έχουμε σαφείς και ξεκάθαρου κανόνε που θα εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση όλων των operators ενώ ο κανόνας θα πρέπει να είναι ο, οι διαγωνισμοί, η πρόταση έχει πολλές εξαιρέσεις για τις άμεσες αναθέσεις, κάτι που μου ζητήθηκε από τον εισηγητή αλλά και από πολλούς ομιλητές. Αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να, περιμένουν, να παραμείνουν περιορισμένες ε, και να χρησιμοποιούνται μόνο όπου είναι απαραίτητο. Το να, δι, διπλασιαστούν ε, ο αριθμό των ε, αναθέσεων που μπορούν, που μπορούν να γίνουν άμεσα, στα 10, να φτάσουν δηλαδή τα 10 εκατομμύρια, δεν θεωρούμε ότι είναι σωστή. Επίση, οι ε, τροπολογίε 27 και 28 ε, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογή τη ε, της πρότασής μας γιατί μιλούν για μετρό και για λεωφορεία, ενώ η δική μας πρόταση μιλάει για σιδηροδρόμους. Η δομή των σιδηροδρόμων και τα χαρακτηριστικά της αγοράς του είναι πολύ, διαφορετικά, πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα και έχουμε και την αρχή της επικουρικότητας που σημαίνει ότι οι περιφερειακές και εθνικές αρχές είναι αυτές που θα ορίσουν τις ανάγκες και θα αποφασίσουν τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για το προσωπικό τους. Τέλος, η, η Κομισιόν προτείνει μια μεταβατική περίοδο μέχρι το 2019 το να αναβληθεί αυτή η περίοδο και να φτάσει το 2029 δεν είναι λογικό. Τροπολογία 31. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι συμβάσεις του, οι άμεσες αναθέσεις που γίνονται μπορούν να γίνουν για μια για χρονική περίοδο 10 ή 15 χρόνων κάτω από ειδικέ συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι άμεσα, ανατιθέμενε συμβάσει μπορούν να συνεχίσουν μέχρι το 2030 ή το 2044 αν δεχτούμε αυτό που προτείνει ο εισηγητή. Μπορούμε να δεχτούμε ότι θα μείνουν κλειστέ οι αγορές για άλλα 20-30 χρόνια. Για το... Γιατί τώρα δρούμε τώρα. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2012-34 ε, απαντά σε μια άμεση έκκληση του κοινοβουλίου σας. Γι' αυτό κλείνοντας θα πω ότι θα πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση αυτής της ε, έκθεσης που θα πάει από τη δική σας επιτροπή στην ε, ΤΡΑΝ. Είναι δική μας ευθύνη να υπάρξει το σωστό πλαίσιο που θα συμβάλλει στην ε, ανταγωνιστική θέση των σιδηροδρόμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Α, ναι, αλλά να σας απανθυμίσω ότι οι πολιτικές αρχές θα καθορίσουν τη γραμμή που θέλουν και όχι η Κομισιόν. Εμείς θα τις υποβάλουμε τη γραμμή. Η Κομισιόν είναι μια τεχνική εμπειρογνωμοσύνη. Κύριε Ισηγητά, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ όσους έλαβαν το λόγο που μίλησαν όχι μόνο για το σχέδιο γνωμοδότησης αλλά και για το θέμα γενικότερα, πλήρως μάλιστα. Διότι δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε ούτε στην ιδεολογία ούτε να θεωρήσουμε ότι το αγγλικό πρότυπο είναι το μόνο και εκείνο που αποδεικνύει ότι χρειάζεται πλήρης απελευθέρωση. Η αντίδραση της Κομισιόν βασιζόταν στη μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζουμε ότι υπάρχει και το θέμα της εγγύησης της προσφοράς στο σύνολο του ενωσιακής επικράτειας καθώς και το θέμα της προστασίας των εργαζομένων, της ασφαλείας και όλα αυτά μέσα στο σωστό χρονοδιάγραμμα. Και Δεν λέω ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν άλλες φάσεις εκτός από εκείνες που αποφασίστηκαν, αλλά νομίζω ότι Πρέπει να επιδείξουμε φρόνηση και να μην αγνοήσουμε πτυχές που ανέφερα πριν, τις πτυχές που ανέφερα πριν. Αλλά θα κάνω ό,τι πρέπει ώστε να συνεννοηθώ με τους κοιόδης για να βελτιωθεί η γνωμοδότηση και να ανταποκρίνεται στην πλειοψηφία εδώ στην Επιτροπή μας. Και φυσικά θα ακούσω με μεγάλη προσοχή τα επιχειρήματα όλων. Ευχαριστούμε κύριε Σιγητά. Η διορία κατάθεσης των τροπολογιών λίγη στις 27 Σεπτεμβρίου με ψηφιακή λέει υπογραφή μέχρι το μεσημέρι. Θα εξεταστούν στις 17 Οκτωβρίου, 14 Νοεμβρίου η ψηφοφορία και ταυτόχρονα στην Επιτροπή Μεταφορών ή μάλλον στις 26 Νοεμβρίου. Τώρα πάμε στο 18 όπου θα δώσω το λόγο στην κυρία Τατιάνα Σδανόκα που θα μας παρουσιάσει τις 24 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί για τη σχέδιο γνωμοδότησής της για την Επιτροπή. Α, όχι, όχι. Α, όχι. Όχι αυτό, εμεί είμαστε αρμόδιοι επί τη ουσία. για τη ενέργεια κλιματολογικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην κοινότητα. Είναι έκθεση για την οποία η, θα γνωμοδοτήσει η Επιτροπή προπολογισμών και 24 τροπολογίες είναι 10 αρχικέ τη εισηγήτρια και 14 υπόλοιπε. Ορίστε κυρία εισηγήτριά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους κοιόδης συζητητές για τις τροπολογίες. Είναι πολύ επικοδομητικές οι τροπολογίες αυτές και θα εμπλουτίσουν την έκθεση. Θα ξεκινήσω με τα εκτιμώντες, με τις τυλικές σκέψεις. Έλαβα μια τροπολογία της Μαλούφου Καστέλου για το εκτιμώντας 1, καινούριο. Και, όπως λέει και η κυρία Κοστέλου, πρόκειται για μια τροπολογία, στη δική μου τροπολογία, ένα συμπεριλαμβανομένης και μια αναφορά στη χάρτα και στο άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Καστελή για την ε, τροπολογία. Και θα καταθέσω μια συμβαστική τροπολογία που θα βασίζεται και σε αυτές τις δύο τροπολογίες. Την 1 και την 11 δηλαδή. Στη συνέχεια, επόμενη τροπολογία αφορά την αιτιολογική σκέψη 3. Εδώ Έχουμε τις τροπολογίες, δύο τροπολογίες, ε, την τροπολογία 12 της Ιδίας και την τροπολογία 13 της κυρίας Χάρκιν. Και για τη συνάντηση των σκιωδών θα προτείνουμε ένα συμβιβασμό. Νομίζω ότι θα είναι δύσκολο να βρούμε μια συμβιβαστική τροπολογία, σε υπόψη και τις δύο αυτές τροπολογίες, 12 και 13. Επόμενη. τροπολογία αφορά το εκτιμώντας 5. Λάβαμε μια τροπολογία. Όχι. Εκτιμώντας 8 διορθώνει μιλήτρια. Η δημιουργική σκέψη 5 ήταν δική μου τροπολογία, αλλά για το εκτιμώντας 8 υπάρχει μια τροπολογία από την Επιτροπή Περιπολογισμών που είναι παρόμοια με μια δική μου, με την υπαριθμόν 3. Έτσι λοιπόν θα είναι εύκολο και εδώ να καταλήξουμε στη συμβαστική τροπολογία. Για να συμπεριλάβουμε και δύο τροπολογίες από δύο σκιώδεις, την κυρία Κοστέλ και την κυρία Χάρκιν. Τροπολογία 14 και τροπολογία 15. αφορούν τη βελτίωση της διατύπωσης. σε σχέση με τη συνεισφορά της Ένωσης ε, και τα Εθνικά Ινστιτούτ Στατιστικών. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμβαστική τροπολογία, λαμβάνοντα υπόψη τι τροπολογίε 14-15, τροπολογία 1 τη Επιτροπή Υπολογισμών και τη δική μου υπαριθμών 3. Για το κτιμώντα 9. Έχουμε και εδώ δύο τροπολογίε από τι ε, ίδιε συναδέλφου. σκεφτούμε το θέμα της διατύπωσης για τους όρους burden ή workload. Πρόκειται για τροπολογίες ε, που αφορούν τη διατύπωση. Η κυρία Καστέλα τα πάει καλύτερα από τα αγγλικά. Επομένως ε, θα καταθέσουμε μια συμβαστική πρόταση. Συμφωνώ ότι κυριε κυριε καστελα τα παει καλυτερα απο τα αγγλικα επομενως θα καταθεσουμε μια συμβαστικη προταση συμφωνω οτι η δικη σας πρόταση είναι καλύτερη από αυτή της Κομισιόν. Έχουμε και την τροπολογία 17 της κυρίας Χάρκιν που αφορά τα διάφορα μοντέλα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες. Και για το σημείο αυτό. Τώρα, άρθρα. Όχι. Έχουμε και την τροπολογία 18 για ένα ακόμα εκτιμώντα το υπαριθμό 12. Και εδώ συμφωνώ. Αφορά κυρίω τη διατύπωση. Πρόκειται για τροπολογία που έρχεται την κυρία Καστέλη. Σύμφωνα απόλυτα λοιπόν με την τροπολογία σα. Τώρα περνάμε στα άρθρα. Έχουμε τη δίκη με τροπολογία για το άρθρο ένα, συζητήθηκε ήδη. Αλλά σε ό,τι φορά τώρα τις τροπολογίες από τους σκιώδεις. Έχουμε τροπολογίες για το άρθρο 1, παράγραφος 2, που αφορά το νέο άρθρο 7β που προτείνεται από την Κομισιόν. Και έχουμε και τις τροπολογίες 19 και 20 έχουμε και την τροπολογία 3 από την Επιτροπή Περιπολογισμών. Νομίζω ότι θα προτείνω συμβαστικές τροπολογίες για τη συνάντηση των σχεδόν συγκητών. Και για τα σημεία αυτά. Βασικά συμφωνώ με αυτές τις προτάσεις. Το ίδιο φορά και στις τροπολογίες 21 και 22 σχετικά με την παράγραφο 2 του άρθρου 7 γάμα που προτείνει η Κομισιόν. Και αυτές είναι καλές τροπολογίες. Θα καταθέσουμε λοιπόν συμβαστικές προτάσεις. Και την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 7 γάμα. Έχουμε μια τροπολογία της κυρίας Χάρκιν, την υπαριθμό 23. Είναι σχεδόν ταυτόσιμη με τη δική μου, υπαριθμό 10. Όταν συζητήσαμε την τροπολογία μου, οι σκιώδεις συμφώνησαν ότι πρέπει να είναι περιορισμένοι στο χρόνο ενώ η κυρία Χάρκιν προτείνει πέντε έτη, μπορούμε να συμφωνήσουμε. Και τέλος, έχουμε την τροπολογία 24. Από την κυρία Σάγια, από το ΕΛΚ. πρόταση της Κομισιόν αφορά και πάλι το 7 παράγραφος 6. Εδώ η Κομισιόν προτείνει δύο μήνες για την κοινοποίηση. Η Εσάγια προτείνει τρεις μήνες. Νομίζω μπορούμε να υποστηρίξουμε και αυτή την τροπολογία. Καλύτερα να έχουμε περισσότερο χρόνο. Αυτά από μένα για αυτές τις τροπολογίες. Και για μια ακόμη φορά ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Euh, ευχαριστώ πολύ για αυτή την εξονυχιστική ανάλυση των τροπολογιών. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Εσαγιά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είχα πει και στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων ότι είμαι ικανοποιημένη από το κείμενο της Επιτροπής, γι' αυτό κατέθεσα μία τροπολογία για την τρίμηνη περίοδο. Και επίσης συμμερίζομαι την άποψη της εισηγήτριας ότι πρέπει να υπάρχει πενταετής περίοδος για την μεταβίβαση των δικαιοδοσιών. Νομίζω ότι το, ελπίζω το συμβιβαστικό κείμενο είναι τέτοιο ώστε να Συμφωνούμε πάντοτε με τη μελέτη για το εργατικό δυναμικό. Αλλά η συγκήτρια εργάστηκε καλά και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και να συνεννοηθούμε. Κοστέλο. Ευχαριστώ κύριε Συγκήτρια και εγώ, ε, κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Συγκήτρια για την εργασία της και να δηλώσω ότι είμαστε υπέρ των ιδεών που μας εξέφρασε για την Ένωση. Οι τροπολογίες που κατέθεσα αφορούσαν τις λεπτομέρειες μάλλον παρά την ουσία αλλά είναι δύο που θα ήθελα να τονίσω η πρώτη είναι η 11 που όπως είπε και η συγγήτρια βασίζεται στη δική της 1 για, αλλά θέλει να υπάρχει μια μεγάλη αναφορά ευρύτερη για τη χάρτα των θεμελιωδών και για το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ένωσης που λέει ότι η Ένωση είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει πλήρη απασχόληση και όχι το 9 που μιλάει απλώς για υψηλό επίπεδο απασχόλησης. Είναι σημαντικές οι διαφορές αυτές. Δεύτερη τροπολογία που θα ήθελα να τονίσω από τις δικές μου είναι η 16. Γιατί εκεί θεωρούμε ότι αν και είναι γλωσσικό μάλλον θέμα, η ιδέα της χρησιμοποίησης του όρου workload είναι καλύτερη από τον όρο administrative burden Γιατί λέμε administrative burden ενώ εννοούμε workload. Όσο για τη στρατηγική 2020 της Ένωσης μπορούμε να κάνουμε εδώ μια παραπομπή για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να μας υποβάλουν στο χρονοδιάγραμμα του 2020. Βέβαια αυτές είναι γλωσσικές όπως είπα και όχι ουσιώδεις. Κατέθεσε και η Μάριον Χάρκιν τροπολογίες με τις οποίες βασικά συμφωνώ. Υπάρχει και 23 για την περιορισμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτό ίσως χρειαστεί να το ξανασυζητήσουμε, αλλά και πάλι ευχαριστώ την εισηγήτρια για όλα όσα έχει κάνει για μας. Ευχαριστώ Χάρκιν και μετά η Κομισιόν που θα εκπροσωπηθεί από το Ευρωστάτ. Η Μαριάννα Χάρκιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δόθηκε από την εισηγήτρια πλήρης ε, περιγραφή των ε, τροπολογιών. Εγώ θα επιτεδοθώ απλώς σε αυτό που λέμε για το διοικητικό άκθος. Ίσως ε, το δυσανάλογο να πρέπει να είναι καλύτερος όρος, δεν ξέρω έχουμε έτσι μια διαφωνία, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε. Και θα συμφωνούσα ότι μπορούμε να λέμε union policies και όχι στόχοι του 2020, γιατί θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο δυνατόν περισσότερα. Και τέλος, για την τροπολογία 20, αυτό που είπατε στο τέλος, για το, η με βάση τη συμμετοχή των κρατών είναι καλό. Και για την 23 μπορούμε να τη συζητήσουμε. Αλλά γενικώ νομίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για το φάκελο αυτό και ευχαριστώ όλους. Ε, Thank you, Chair. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Yes, I must catch a train, me too, to Luxembourg. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την εισηγήτρια και τους σκιώδες για τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της πρώτης κομισιόν. Δύο πράγματα θα πω. Το πρώτο είναι το αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν εφαρμοστικά μέτρα ή κατεξοδότηση πράξης. Εδώ να πω ότι η Κομισιόν πιστεύει ότι τα εφαρμοστικά μέτρα είναι πιο κατάλληλα όταν πρόκειται για τεχνικά θέματα, όπως αυτό εδώ. Ε, μιλούμε για ένα θέμα τεχνικής φύσεως, αυτό που συζητούμε εδώ. Οπότε, η πρόταση της Κομισιόν είναι να υπάρχουν εφαρμοστικά μέτρα για τα τεχνικά σημεία. Δεύτερον, η χρήση των καταποκοπή ποσών για, τα, για την επιδότηση στα κράτη-μέλη. Ε, αν θα λέμε may ή will μέσα στην πρόταση. Είναι καλύτερο να είναι καταποκοπή πληρωμές, καταποκοπή ποσά οι πληρωμές ε, και να το κάνουμε κάπως υποχρεωτικό αυτό. Εμείς θέλουμε να υπάρχουν απλοποιημένες δικασίες για, την, ε, για τις επιχορηγήσεις. Οπότε θεωρούμε ότι το may μπορεί είναι ίσως πιο ευέλικτος όρος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτές τις τεχνικές διευκρινήσεις. Να ξαναδώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ τους και τους Σα Σας ευχαριστώ που υποστηρίζετε τη θέση μου. Θα τα συζητήσουμε και στη συνάντηση των σχεδόν συγητών και κατά τη διάρκεια των τριμερών διαλόγων θα συζητήσουμε τα ευαίσθητα θέματα των κατεξουσιοδότηση πράξεων, των θεριστικών πράξεων κτλ. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πάντα πρόβλημα, αλλά θα βάλουμε τα δυνατά μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε τις θα συζητήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες στην επόμενη συνεδρίαση. Όχι στις 17 Οκτωβρίου και θα τις υιοθετήσουμε εγκαίρως για να μπορέσουμε να πάμε στη Ρωμέλη όταν θα έχουμε μία κοινή θέση. Με το Συμβούλιο ολοκληρώσαμε και αυτό το σημείο στην διάταξη. Το σημείο 10 θα δώσω το λόγο στην Φρασουάζ Καστέξ για να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της και να τοποθετηθεί επί τροπολογιών που κατατέθηκαν στη γνωμοδότηση σχετικά με την ετήσια έκθεση, σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μία έκθεση πρωτοβουλίας ε, όπου ο κύριος Τρεμός Έμπαλτσετς είναι ο εισηγητής στην Επιτροπή κυρία Κύριε Καστέξ, ευχαριστώ. Έχω κάποιες συμπληρωματικές τροπολογίες για το σχέδιο γνωμοδότησης από τους κύριους Κάζα, Καστέξ, Κλειβέτη, και άλλους και διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι αυτές οι τροπολογίες πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση με τη δική μου γνωμοδότηση. Δηλαδή, ότι η πολιτική ανταγωνισμού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ρόλο που της έχει αποδοθεί από τις ε, συνθήκες, δηλαδή από το να προστατεύει τον καταναλωτή από τις αθέμητες πρακτικές ε, και να σταθεροποιεί την εσωτερική αγορά, όμως ε, υπήρχε ουσιαστικά μία παρέκκληση στην πολιτική ανταγωνισμού όταν εκεί μιλούσαμε για χρηματοδότηση δημοσίων επιχειρήσεων και για κρατικές επιδοτήσεις και μάλιστα και στην τελευταία έκθεση της ε, Επιτροπής Ανταγωνισμού γίνεται λόγος για μια πολιτική η οποία εξυπηρετεί την λιτότητα. Δεν ήταν λοιπόν πολύ δύσκολο να προτείνω στους συναδέλφους μου συμβαστικές τροπολογίες. Πρότεινα 7-8 που έγιναν αποδεκτές. παραμένει μια τροπολογία που θα πρέπει κάπως να διορθωθεί. Αφορά μια από τις συμπληρωματικές μου τροπολογίες, τη 43, τη 42 της κυρίας Ρέκνερ, την 24 της κυρίας Κλιβέτη και άλλη μια τροπολογία όπου Θέλουμε να υπενθυμίζουμε ότι είναι και ρόλος της Κομισιόν να περιορίσει τις ε, πρακτικές όπως είναι το κοινωνικό dumping και το φορολογικό dumping, αντικοινωνικές δηλαδή πρακτικές. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πρέπει να διατυπώσουμε και τις λεπτομέρειες. Η κυρία Ρέκνερ, μάλιστα, έχει απαριθμίσει όλα τα στοιχεία στρέβλωσης και ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών, ε, δηλαδή τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας, ε, τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, το φορό των επιχειρήσεων και τα μέτρα καταπολέμησης της ε, φοροδιαφυγής και της φοροπάτης. Ενώ σε άλλη περίπτωση αποφεύγεται η απαρίθμηση τόσο συγκεκριμένων στοιχείων. Στην άλλη τροπολογία του συναδέλφου. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να βρω μια διατύπωση με την οποία όλοι είναι σύμφωνοι και να μπορέσει να ψηφιστεί αυτή η γνωμοδότηση από την Επιτροπή Απασχόλησης και να μπορέσουμε να διαβιβάσουμε στην Επιτροπή ΕΚΟΝ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού μια γνωμοδότηση δική μας ε, της Επιτροπής Απασχόλησης που θα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι η πολιτική ανταγωνισμού παραμένει εκεί που είναι και δεν επηρεάζει τις πολιτικές κρατικών ενισχύσεων, τις κοινωνικές πολιτικές και των δημόσιων υπηρεσιών. Euh, euh, Η κυρία Ρόιτεν που αντικαθιστά το σχεδόν συγγητή του ΕΛΚ. Ε, ε, First... Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ εκ μέρους του κυρίου Κάζα την κυρία Καστέξη για τη δουλειά που έκανε. Ο Ντέιβιντ μου είπε ότι το αρχικό σχέδιο της έκθεσής της ήταν πολύ καλό, ισορροπημένο και μπορεί να υποστηρίξει τις περισσότερες από τις τροπολογίες. Το πρώτο σχέδιο των τροπολογιών, όπως είπατε, ήδη έχει κυκλοφορήσει. Ο κύριος Κάζα ήθελε κάποιες ε, διευκρινήσεις για τις συμβαστικές τροπολογίες, αλλά ήδη είπε ότι μπορεί να συμφωνήσει με τα περισσότερα από τα θέματα. Όπως είπατε και περιμένει και ο ίδιος ε, το τελικό χτένισμα των τροπολογιών τις επόμενες μέρες. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρξει ε, συμφωνία, θεωρεί ο ίδιος και σα ευχαριστώ εξ του. Ευχαριστώ. Θέλει άλλο το λόγο. Μπερδεύτηκα λίγο στην αρχή με τις, γιατί δεν κατάλαβα, συζητούσα με τις συμβαστικές και τις τροπολογίες. Πρώτη φορά συζητούμε τις τροπολογίες σήμερα. Αλλά ήδη φτάσαμε στις ε, συμβαστικές τροπολογίες, οπότε μάλλον το πρώτο θέμα ελήθη. Λοιπόν, για τις τροπολογίες έχουμε τέσσερις που βρίσκονται στο, αφορούν μάλλον στο ίδιο σημείο, την εξασφάλιση, ε, της συνεχτικότητας, της, της πολιτικής ανταγωνισμού, σε ό,τι αφορά τους κοινωνικούς, οικονομικούς ε, και περιβαλλοντικούς στόχους. Έχω επιβάλει αρκετές τροπολογίες ως προς αυτό. Επίσης υπέβαλα μια τροπολογία που δεν υποστηρίζει πλήρως την παράγραφο 5 και προέδινα και ένα εναλλακτικό κείμενο για την παράγραφο 5. Και από τις αρχικές τροπολογίες, οι δύο της κυρίας Κορνέλισεν για το level playing field, η τροπολογία 4 του εισηγητή και η 19 της κυρίας Καστέλο που έχει να κάνει με την ε, εκπαίδευση και την κατάρτιση μπορούν να γίνουν αποδεκτές από μένα. Έχω κάποιες ανησυχίες για τις τροπολογίες που δημιουργούν πολλές εξαιρέσεις, που σημαίνει ανισορροπία στην αγορά και άρα υπονόμευση της όλης πολιτικής. Γενικώ όμως, ε, είμαστε ικανοποιημένοι με τις περισσότερες από αυτές και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές προτάσεις. Τώρα, για τις συμβαστικές προτάσεις, Έχω έτσι κάποιους συνδυασμούς για πολύ μικρά κομμάτια της διατύπωσης. Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο σπαστικός με αυτό, αλλά τέλος πάντων έχω κάποιες αντιρρήσεις με τη διατύπωση. Προφανώς το μακροπρόθεσμο είναι καλύτερο από το βραχυπρόθεσμο. Το unable που λέει μέσα στο κείμενο δεν είναι σωστό. Θα πρέπει να λέμε ότι δεν είναι δυνατόν να το ανίκανο είναι λίγο ισχυρή λέξη. Για το G, αντί να λέμε ειδικός, ειδική δέσμη κανόνων, αλλά λέμε ευελιξία εντός του τρέχοντος πλαισίου κανόνων. Αν αρχίσουμε να βάζουμε διάφορους, διάφορες δέσμες κανόνων, θα γίνουν τα πράγματα πολύ περίπλοκα. Ε, βεβαίως, ε, παραδέχομαι ότι χρειάζεται κάποια ευελιξία. Για, την για τη συμβαστική H συμφωνούμε ότι ε, ο διάλογος δεν θα πρέπει να, που προτείνει η Κομισιόν δεν θα πρέπει να αντικαθιστά τον δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου. Βεβαίω ο διάλογος πρέπει να παίξει τον ρόλο που του αναλογεί στην ε, ε, πολιτική ανταγωνισμού και στα πλαίσια των ευρωπαϊκών και εθνικών προτεραιοτήτων. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Αυτά από μένα. Αυτά ήταν τα σχολιά μου. Ε, merci. Est-ce Θέλει κάποιος άλλος το λόγο, όχι. Να προτείνω στη διαπραγματευτική ομάδα και εγώ κάτι. Κάπως καθυστερημένα βέβαια, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια παραπομπή στο άρθρο 14 της συνθήκης του πρωτοκόλου για τις δημοσίες υπηρεσίες ε, και ξέρετε ότι εμείς πάντα ως Επιτροπή Απασχόλησης ε, πάντοτε έχουμε συμφέρον υπερθυμίζουμε τη μάχη που δώσαμε για να εγγραφεί το άρθρο 9 στη συνθήκη που επιτρέπει να δηλώνουμε και την πολιτική ανταγωνισμού. Τελικά δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί διαμάχες μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν, ε, ίσως ε, θα μπορούσατε να προσθέσετε μια σχετική παραπομπή. Ίσως είναι αργά που το θέτω, αλλά σκέφτηκα ότι ίσως ε, θα έπρεπε να έχει τεθεί και το θέμα αυτών των ε, μεγάλων δομών Amazon, Google, ε, Facebook, Apple που μέσω διάφορων φορολογικών στρατηγικών οδηγούν σε μετακίνηση των θέσεων εργασίας και η Κομισιόν ε, δεν λέει τίποτα σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό. Μια προφορική τροπολογία για το άρθρο 9 νομίζω ότι δεν θα έφερε πρόβλημα και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε να στέλνουμε το μήνυμα αυτής της Επιτροπής. Δεν ζητά άλλο το λόγο, να ξαναδώσω το λόγο στην συγγήτρια. Πρόεδρε, Πράγματι δεν ε, ανέφερα εγώ το άρθρο 9 στην αρχική μου γνωμοδότηση, αλλά θα κάνω αυτή την παραπομπή, καθώς ε, θα θετήσω και μια τροπολογία του κυρίου Σέρκα, στην υπερθυμόν 21. Και προφανώς ε, θα ψηφιστεί. Ζητώ συγγνώμη από το κύριο Μπενιόν. Έλαβα υπόψη τις ε, τροπολογίες του σε δύο συμβαστικές προτάσεις, ε, στην 33 και στην 39 τροπολογίες που ανέφερε. Τώρα για τους συμβιβασμούς E και H θα αναφερθεί και σημασία του κοινωνικού διαλόγου και η σημασία του δημοκρατικού ελέγχου του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι και για αυτά τα θέματα υπάρχει, διαφαίνεται μια συνένεση, γιατί σήμερα μόνο η Κομισιόν έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την Επιτροπή για την πολιτική, με συγχωρείτε, ανταγωνισμού και αυτό αμφισβητείται. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εξαιρέσεις που προτείνονται για την πολιτική ανταγωνισμού, αφορούν μία ελάφρυνση του βάρους του ανταγωνισμού στις κρατικές ενισχύσεις, δηλαδή για τη δημόσια παρέμβαση στην οικονομία για να δοθεί νέα όθηση στη βιομηχανία. Είχαμε μια σχετική τροπολογία από τον κύριο Μπουλάν και για την προστασία των κοινωνικών πολιτικών και των δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης υπάρχει μια εξαίρεση με ελάφρυνση της πολιτικής ανταγωνισμού που προτείνω εγώ για την δομή της ε, κοινωνικής, για τις δομές της κοινωνικής οικονομίας. το χάρη, τα ταμεία βοήθειας, ε, τις κοπερατίβες και δεν θα έπρεπε οι δομές αυτές ε, να την χάνουν ίδιας μεταχείρισης όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές είναι οι μόνες εξαιρέσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στην πολιτική ανταγωνισμού. Θα συνεχίσω να μελετώ τις συμβαστικές προτάσεις και να τις επεξεργάζομαι και εγώ νομίζω ότι τώρα είναι απλώς θέμα διατύπωσης, δεν νομίζω ότι έχουμε προβλήματα ουσίας και δεν αμφιβάλλω ότι αυτή τη γνωμοδότηση θα μπορέσουμε να την ψηφίσουμε με μεγάλη ομοφωνία. Ευχαριστώ. Ε, Στη βάση αυτού του συμβιβασμού που θα εκπονήσετε, θα εξετάσουμε στις τροπολογίες στις 25 Σεπτεμβρίου, την επόμενη συνεδρίασή μας λοιπόν, και θα ψηφίσουμε την επόμενη ημέρα. Και η Επιτροπή Οκών θα ψηφίσει στις 17 Οκτωβρίου. Τώρα φτάνουμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης και το λόγο θα πάρει η συγγήτρια η κυρία Σαρτιέ για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Απλώς ε, θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι αμέσως μετά τη συνεδρίασή μας θα λάβει η χώρα ο 26ος τριμερής διάλογος και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και ακόμη τριμερούς διαλόγους. Πρέπει όμως να πω ότι καταρχήν αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να διατηρήσουμε όλες τις κοινωνικές πολιτικές που είναι πολύ σημαντικές για αυτή την Επιτροπή. Είχαμε μια εντολή πολύ ισχυρή στο βαθμό που στη δική μας Επιτροπή υπήρχε μεγάλη συνοχή μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και αυτός ε, είναι ο δεύτερος λόγος για τον οποίο έπρεπε να αναλάβουμε αυτούς τους πολύ βαρύς διαλόγους είναι ότι η πρωτοβουλία για την απασχολησιμότητα των ε, νέων ήρθε να προστεθεί σε ένα πρόγραμμα διαπραγματεύσεων ήδη αρκετά βαρύ. Τώρα, για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Να σας δώσω κάποιες πληροφορίες ε, που δεν ε, ήταν βέβαιες, αλλά έλαβα μία επιβεβαίωση. Υπάρχουν επιστώσεις σε front-loading που έχουν γραφεί για τον προϋπολογισμό 2014 για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των Θυμάστε ότι είχαμε κάποια αμφιβολία. Υπάρχουν πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, 6 δισεκατομμύρια ευρώ Νομίζω ότι μιλάμε για 1,8 ε, δισεκατομμύρια και κατόπιν πιστώσεις ε, πληρωμών. Ναι, ε, ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολλά τα χρήματα, αλλά γι' αυτό ακριβώ υπήρχε αυτός ο φόβος. Όμως, σύμφωνα με όσα μου λένε, αυτό αιτιολογείται από το γεγονό ότι πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά. Δηλαδή, έχουμε μία απάντηση στην ανησυχία μας, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει διασκεδαστεί εντελώς η ανησυχία μας. Και κάτι ακόμη για τις διαπραγματεύσεις, τις οποίες βρισκόμαστε. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε ένα άνοιγμα ε, προς ε, το, ε, την ηλικία μέχρι τα 30, την ομάδα αυτή την ηλικιακή, για τους νέους ανέργους από 15 έως 25 έτη. Με συγχωρείτε. Ναι, μέχρι τα 25 αυτό είναι. Δεύτερον, θα θυμάστε ότι εμείς θέλαμε να λάβουμε υπόψη και τις περιφέρειες όπου ε, έχουμε πάνω από 20% άνεργους νέους ε, σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Και αφού συζητήσαμε με την Κομισιόν, είδαμε ότι ο Ευρωπαϊκός Μέσος Όρος ήταν 22,9 το 2012 και 22,8 το 2013. Ναι. Και μελετήσαμε αυτό τον ε, ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν ε, δηλαδή λαμβάνουμε υπόψη αυτό τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε το πεδίο εφαρμογής ε, και τελικά περάσαμε στις 121 ε, περιφέρειες και μία και μόνη χώρα θα υποφεληθεί από το 1 τρίτο αυτής της αύξησης. Επομένως συνεχίζουμε τις συζητήσεις αυτές. νομίζω ότι σας ανέφερα τα κυρία σημεία τα οποία συζητούμε σήμερα και την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Γνωρίζοντας βέβαια ότι τίποτα δεν έχει σταθεροποιηθεί μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κερδίσει σε κάτι σήμερα περισσότερο από σε κάτι άλλο, γιατί είναι καθολικές οι διαπραγματεύσεις. Και όλες οι προεδρίες άνοιξαν όλα τα συρτάρια αλλά δεν τακτοποίησαν κανένα. Bien, euh, θέλει κανείς να πει τίποτε συμπληρωματικό. Τα αποτελέσματα του τριμερούς διαλόγου θα τα έχετε το βράδυ και θα συζητηθούν στην επόμενη μας συνεδρίαση στις 23-25 Σεπτεμβρίου στις 3 με κύριο θέμα το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο ως παράγοντα ανταγωνιστικότητας σε συνεργασία με τις τέσσερις υπηρεσίες. Και μετά θα συνεχίσουμε τα κανονικά το απόγευμα στις 25 και στις 26 το πρωί. Καλή νύχτα.